πάρα πολύ κύριε Επιτροπέ. 14 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Υπόδειγμα για όλους. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο να δούμε αν θα μπορέσει να σας μιμηθεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, συγχαρητήρια για την ε, υποψηφιότητα αυτή και το διορισμό σας. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις ε, ικανότητές σας και τις δεσμεύσεις σας εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε περάσει τα πειρά μια τέτοια ακρόαση και πριν από πενταετία και έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά ω Επίτροπο Περιφερειακή Πολιτική ήδη. Να θυμίσω κάτι που και στην συνάντηση τη περασμένη εβδομάδα αναφέρατε. Είπατε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε το συνήθειο να μπαίνετε ω μπουλντόζα στην καρδιά των προβλημάτων για να τα συζητήσετε. Αυτό προκάλεσε πολλά σχόλια διότι αυτό στην επιστολή με τις αρμοδιότητές σας είναι σημαντικό. Πιστεύετε ότι θα έχετε περισσότερες αρμοδιότητες από τον Επίτροπο που θα είναι επιφορτισμένος με θέματα διεύρυνσης. Και τα δύο. Μπορώ να σας απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα για να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Και τα δύο. Je suis totalement satisfait. Ε, είμαι πλήρως ε, ικανοποιημένος. Ο κύριος Χόουιτ. Στον τίτλο των αρμοδιοτήτων σας υπάρχει ο όρος διεύρυνση. Με τις διαπραγματεύσεις όμως τι θα γίνει. Θα ήσασταν επίτροπος διεύρυνσης και, περιφερειακής, ε, και πολιτικής μάλλον γειτονίας. Θα ήταν μια αλλαγή που θα μπορούσατε να δεχτείτε. Επίσης, εάν δεν υπάρξουν περαιτέρω διευρύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την επόμενη πενταετία. Ποια θα είναι τα κριτήρια επιτυχίας που θα έχετε θέσει στον εαυτό σας για την ε, ε, ευρωπαϊκή πολιτική διεύρυνση στη δική σας θητεία. Επίσης, στην Αυστρία υπάρχει μικρότερη στήριξη για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο σας ε, ένα δείγμα ότι υπάρχει κόποση στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχει φτάσει αυτό και στις Βρυξέλλες και πώ θα φροντίσετε από τις Βρυξέλλε να αλλάξει κοινή γνώμη ω προς αυτά ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην περασμένη σας θητεία ως ε, Επίτροπος, πόσον καιρό έπρεπε να περιμένετε με υπομονή για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και ε, πόσο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να προσπαθήσετε πριν εγκαταλείψετε κάποια προσπάθεια, εφόσον θα υπάρχει ένα ολόκληρο σώμα να πιστεί. Για την πρώτη σας ερώτηση. Δεν υπάρχει αντίφαση. Είναι σαφές όσο πρέπει να εστιάσουμε στις ε, διαπραγματεύσεις της διεύρυνσης και όπως είπα το θέμα είναι η ποιότητα και όχι η ταχύτητα. Εγώ έχω μεγάλη εμπειρία από τα καθήκοντά μου ως Επιτροπός Περιφερειακής Πολιτικής και είναι προς το συμφέρον μας να είναι προετοιμασμένα τα νέα κράτη-μέλη και έτοιμα να εφαρμόσουν ε, και να εκμεταλλευτούν όλες τις ευκαιρίες που έχουν π.χ. τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς κτλ. Γι' αυτό νομίζω λογικό είναι να έχουμε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας. Και ακριβώς το ζήτημα είναι να προετοιμάζουμε καλά την, ε, τις μελλοντικέ διευρύνσεις. Για την κοινή γνώμη πράγματι είναι κάτι που πρέπει να δούμε και στα κράτη-μέλη μας. Το θέμα δεν είναι μόνο να διαπραγματευόμαστε με τους εταίρους μας για τη μελλοντική ένταξη, αλλά πρέπει να πείσουμε και τους λαούς μας για τα ωφέλη της μελλοντική διεύρυνσης και για αυτούς, για την ανάπτυξη, τις δουλειές στα κράτη-μέλη γιατί αν δείτε ποιες είναι οι ανερχόμενες ε, αγορές στην Ευρώπη, είναι στην Ανατολική Ευρώπη, οπότε είναι λογικό να επενδύσουμε. Τέλος, να σας διαβεβαιώσω πως είμαι αρκετά υπομονετικός. Θα είμαι στη δουλειά μου, δεν δουλεύω 8 με 5, θα δουλεύω όλη μέρα και τα Σαββατοκύριακα αν χρειάζεται για να πετύχω τους στόχους μας. it? no, that's the... yeah. Σας ευχαριστώ. για αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχει αντίφαση για την υπομονή εγώ φοβάμαι μη φύγει ο συνομιλητής μας από το τραπέζι παρά εσείς για την ποιότητα που μιλήσατε και όχι την ταχύτητα στέλνετε ένα μήνυμα στους ε, συνομιλητές μας στις υποψήφιες χώρες. Ε, μήπως ε, θέλετε να στείλετε αυτό το μήνυμα και μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Κοιτάξτε. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Θα πάω στις χώρες αυτές μόλις αναλάβω τα καθήκοντά μου για να ξεκαθαρίσω πως ε, είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τις ε, σκληρές ε, και επίπονες αυτές διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχία στα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χάν, ως Επίτροπος θα ασχοληθείτε και με τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και υποθέτω πως θα εφαρμόσετε με τρόπο αυστηρό τα κριτήρια. Σε αυτά τα κριτήρια αναφέρεται πως η Τουρκία είναι ένας παράγων σταθερότητας στην περιοχή. Αυτό όμως δεν ισχύει. Βλέπουμε τεταμένες σχέσεις με το Ισραήλ που είναι μάλλον ο μόνος παράγοντας σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Κύριε υποψήφιοι Επίτροπε, ποιο... πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο της Τουρκίας στην Μέση Ανατολή και τι σκοπεύετε να κάνετε για να βελτιωθούν οι σχέσεις ε, Τουρκίας και Ισραήλ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι εν γέννη θα συζητήσουμε το θέμα αυτό αρκετά συχνά γιατί είναι σημαντικό να δούμε την Τουρκία σαν έναν σημαντικό εταίρο για την Ευρώπη και θα πρέπει να έχουμε ένα ενδιαφέρον να βελτιώσουμε και να εμβαθύνουμε στη σχέση μας με την ε, Τουρκία. Και βεβαίως με το θέμα αυτό θα ασχοληθώ ιδιαίτερως και θα δουλέψω εντατικά. Και βεβαίως έχουμε και ένα ενδιαφέρον στην άμεση γειτονία μας να δημιουργήσουμε μια σταθερή και ειρηνική ε, κατάσταση. Και αυτό περιλαμβάνει βεβαίως τις σχέσεις των γειτόνων μας μεταξύ τους. Και υπό την έννοια αυτή και εφόσον είναι αναγκαίο, εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένος, αλλά ασφαλώς και η ύπατη εκπρόσωπος να διαμεσολαβήσει και να εξασφαλίσει ούτε ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης τα κριτήρια ένταξης ανήκει η προστασία και ο σεβασμός των μειονοτήτων στις υποψήφιες χώρες. Πώς κρίνεται λοιπόν τη σημερινή θέση της μικροσκοπικής ε, Ιουδαϊκής και Χριστιανικής κοινότητας στην Τουρκία και σκοπεύετε να κάνετε κάποιες παραστάσεις για αυτά τα θέματα στις ε, τουρκικές αρχές. Ε, σκέφτομαι εδώ πέρα επίσης τα τρομακτικά γεγονότα που είχαμε όσον αφορά την μικροσκοπική, όπως είπα, εναπομείνασα Ιουδαϊκή κοινότητα στην Τουρκία. Έχετε δίκιο και πραγματικά αυτή είναι μια από τις βασικές ανησυχίες που έχουμε με την Τουρκία. Και αν οι ενταξιακές διαπραγματεύσει ε, θα πρέπει να επισπευτούν. Είναι αναγκαίο βεβαίως ε, η Τουρκία και οι πολιτικά ηθήνοντες να κινητοποιηθούν, όχι μόνο να κινητοποιηθούν σε διάφορους τομείς, αλλά και να αποδείξουν ότι πραγματικά παίρνουν σοβαρά τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, κύριε Χάν, θα έχετε τρία αφεντικά. Την κυρία Μογκερίνη, τον κύριο Τίμερμαντ και τον κύριο Γιούνκερ ίσως και περισσότερους. Πώς θα λειτουργήσετε σε αυτή τη νέα δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι εργαστήκατε και στην παλαιά Επιτροπή και θα είσαστε τώρα στη νέα. Τι θα κάνετε όταν σας δίνει κατευθυντήριες γραμμές η κυρία Μογκερίνη. Δεύτερη ερώτηση. Τα λόγια του κυρίου Γιούνκερ. Καμία διεύρυνση. Είναι αυτό ένας λόγος κενός νοήματος διότι αν μια χώρα είναι έτοιμη θα πρέπει να μπορεί να προσχωρήσει. Αυτός είναι ο κανόνας. Και τελευταία παρατήρηση, η ομάδα μου, η ομάδα των φιλελευθέρων, ήταν ε, φυσικά κατά της ρωσικής επίθεσης και εισβολής στην Ουκρανία, αλλά θα πρέπει να έχει και ένα σχέδιο για την στρατιωτική της ακαιρεότητα, ένα σχέδιο Μάρσαλ ουσιαστικά η Ουκρανία για την οικονομική της ανάπτυξη και τη δημοκρατική της σταθερότητα. Παρακαλώ απαντήστε μου. Θα είναι λίγο δύσκολο να σας απαντήσω για το μέλλον της Ουκρανίας σε ένα μισή λεπτό. Πρώτα απ' όλα για την συνεργασία. Δεν ανησυχώ ότι θα τα καταφέρουμε και στην προηγούμενη Επιτροπή. Πολλές φορές έχουμε προσκληθεί να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Δεν βλέπω να δημιουργούνται νέα εμπόδια των αντίον. Το γεγονός ότι τώρα κάποιος από τους αντιπροέδρους θα ασχολείται με ένα θεματικό κλάστερ, ένα σύνολο θεμάτων, σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάποιοι γενικοί βασικοί στόχοι στην Επιτροπή Juncker. Και αυτό είναι σεβαστό από όλου μας. Η δήλωση καμιά διεύρυνση, νομίζω το έχουμε εξηγήσει ήδη, αφορά την ολοκλήρωση και τη σωστή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Φέτος ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο. Εάν δείτε τη διάρκεια που προβλέπετε, μπορούμε να φανταστούμε ότι θα ολοκληρωθούν κάποιες διαπραγματεύσεις γρήγορα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια προθεσμία που πρέπει να τηρηθεί. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι όχι απλώς να συμφωνηθούν όλα σωστά, να συμφωνηθούν εφόσον υπάρξει βελτίωση όντως της επιδόσης των χωρών στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διαφάνεια, στην ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου, Ξεπέρασα νομίζω το χρονικό όριο. Σε μια άλλη ευκαιρία θα μπορούσα να σας εξηγήσω για την Ουκρανία. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω την ε, ερώτηση για την Ουκρανία και να ζητήσω να μου απαντήσετε. Ωραία. Και εδώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια στενή συνεργασία όχι μόνο με όρους πολιτικής, αλλά και για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση της Ουκρανίας, ούτως ώστε να εφαρμόσει όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Δεν πρόκειται μόνο... Ε, το θέμα δεν είναι πάντοτε τα χρήματα, αλλά πάντοτε, αλλά ε, ε, ενίοτε το ζητούμενο είναι να δώσουμε την ε, συνδρομή μας. Και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να βοηθήσουν την Ουκρανία όσον αφορά την αποκέντρωση ή την περιφοριοποίηση της πολιτικής. Επίση, ένα άλλο ζητούμενο είναι η σταθεροποίηση της κοινωνίας των πολιτών καθώς και η ανασυγκρότηση της Ανατολικής Ουκρανίας, όπου βεβαίως ασφαλώς θα χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε εκεί και τα εργαλεία που διαθέτουμε, αλλά όχι μόνον με στενά οικονομικούς όρους. κύριε Χάν, όσον αφορά τη μελλοντική πολιτική γειτονίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, ε, στο υπόβαθρο ότι στο παρελθόν οι συμφωνίες εταιρική σχέσης και σύνδεσης ε, αφορούσαν κυρίως επαναπρόθεση των ε, μεταναστών ή μάλλον περιλάμβαναν κάποια τέτοια στοιχεία και ε, υπάρχουν ε, έτσι διάφορες ε, ευκαιρίες για τις τοπικές ελίτ αλλά και προβλήματα μαζικής εξαθλίωσης σε αυτές τις χώρες. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα πώς θέλετε να προσεγγίσετε αυτά τα προβλήματα με τη βοήθεια της πολιτικής γειτονίας και ποια είναι τα βασικά στοιχεία μιας κοινωνικά δίκαιης και βιώσιμης πολιτικής γειτονίας. Κυρία Λόζινγκ, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να θυμηθούμε εδώ ότι δεν ε, υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλες τις χώρες, αλλά θα πρέπει να δούμε ξεχωριστά τι συμβαίνει σε κάθε χώρα και να αξιολογήσουμε ε, ανάλογα με το επίπεδο προόδου ε, τα μέτρα που θέλουμε να λάβουμε. Γιατί αν δούμε τι γίνεται στην Τινησία και στο Μαρόκο, εκεί έχουν γίνει ε, σημαντικές πρόοδοι. Απ' την άλλη, αν πάρουμε τη Λιβύη, ε, από εκεί το πιο πήγον είναι ε, απλούστατα να εξασφαλίσουμε συνθήκες ασφάλειας για τους πολίτες της χώρας αυτής. Και σε ένα δεύτερο βήμα να εξασφαλίσουμε να λειτουργούν τα εντελώς βασικά για την επιβίωση, δηλαδή να μπορούν οι άνθρωποι να διαβιούν και να εργάζονται με συνθήκες ασφάλειας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ξεχωριστά ατομικά ε, τι συμβαίνει στην κάθε χώρα και να εξασφαλίσουμε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι απολύτως βασικό. Και η εμπειρία μας μας δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι ε, ζουν ε, σε συνθήκες ανεξαρτησίας και ελευθερίας χωρίς φόβο, τότε μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα πράγματα και ε, όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Και ακριβώς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί, κινηθούν οι προσπάθειές μας εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ταυτόχρονα παροχή βοήθειας προς χώρες αυτές ούτως ώστε να εξελιχθούν και να γίνουν οικονομικά αυτοτελείς. Συγκεκριμένα με την κρίση στην Συρία, στις ε, χώρες στις οποίες καταφεύγουν οι άνθρωποι, Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο, υπάρχουν παραβιάσεις ε, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και δεν μπορούν να αποκτήσουν π.χ. το καθεστώς του πρόσφυγα ή να πάνε τα παιδιά του σχολείο κτλ. Τι ε, σκέφτεστε να κάνετε για να χρησιμοποιήσετε την πολιτική γειτονίας ε, και τις αντιπροσωπείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσετε τα, την κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Κοιτάξτε, ναι, το σημαντικότερο είναι να υπάρξει μια ειρήνευση πρώτα απ' όλα στην σύγκρουση αυτή, γιατί πράγματι είναι η κατάσταση δραματική και έχει λάβει γιγάντιες διαστάσεις. Το 2014 είχαμε περισσότερους πρόσφυγες από ότι το 1945. Πότε δεν είχαμε τόσους πολλούς πρόσφυγες ε, παγκοσμίω ε, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν οι βασικές υποδομές γιατί έρχεται και χειμώνας ε, που και σε αυτές τις χώρες είναι βαρύς. Να υπάρχει πρώτα απ' όλα μια διαμονή και ως επόμενο βήμα πράγματι δυνατότητες για τα παιδιά να πάνε σχολείο να μην ε, διακοπεί η εκπαίδευσή τους αλλά ε, όλα αυτά εξαρτώνται και από την ειρήνη και χωρίς μια λύση της σύγκρουσης εκεί πέρα το πρόβλημα των ε, προσφύγων με τις τραγικές πτυχές του δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Μέζεριτς, ε, σας ευχαριστώ κύριε Χάν για τη σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίασή σας. Χάρηκα που άκουσα ε, ότι τονίσατε πως ε, όταν είχαμε επινοήσει την πολιτική γειτονία κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τεράστια κρίση που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ θα έλεγα την ανατολική πολιτική γειτονία θα τη χαρακτήριζα το πολύ μισή επιτυχία. Δηλαδή οι χώρες με τις οποίες έχουμε εταιρική σχέση είναι υποκατοχή, αρκετές από αυτές. Μήπως θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε σοβαρά λοιπόν την ανατολική εταιρική σχέση και ποιος θα συμμετέχει σε αυτήν και άλλη μια ερώτηση. Είδαμε την αρχή της ευελιξίας που αναφέρατε και αυτό ήταν θετικό. Πώς είναι απλά η αρχή περισσότερα έναντι περισσότερων. Εμείς συζητάμε και αρχή λιγότερα με λιγότερα ανταλλάγματα. Γιατί βλέπουμε πως η άλλη τακτική δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, ειδικά στην νότια γειτονιά μας. Νομίζω οι δύο ερωτήσεις συνδυάζονται. Εάν δείτε την επιστολή για την θητεία μου, αυτή που μου απέστειλε, που μου έδωσε ο πρόεδρος Μπαρόζο, ε, μου ζήτησε μέσα σε ένα χρόνο από τη στιγμή που θα αναλάμβανα τα καθήκοντά μου να υποβάλω πρόταση για μια μεταρρυθμισμένη νέα πολιτική γειτονία. Κάτι που θα συμπεριλάμβανε όλα αυτά τα σχόλια, τις αποκρίσεις, τις δικές σας, τους δικούς σας προβληματισμούς. Περισσότερα για περισσότερα ή λιγότερα για λιγότερα και την ανάλογη αρχή. Στο παρελθόν δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στο more for more, περισσότερα για περισσότερα. Αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και όλες τις ευκαιρίες που έχουμε στη διαθέσή μας, όχι για να επιβάλλονται κυρώσεις, αλλά για να δούμε και τη διάσταση λιγότερα για λιγότερα με τον ευστοχότερο τρόπο. Όμως, βασική μας μέρημνα θα πρέπει να είναι να συνδράμουμε τις χώρες αυτές, να τις στηρίξουμε, αλλά είναι δική τους ε, η ευθύνη, του λαού τους, το, κατά πόσον θα κάνουν κυρίαρχες επιλογές για το δικό τους το μέλλον. Βλέπουμε οι χώρες να αποφασίζουν και για τον εαυτό τους και αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Yeah? No. Then uh, Lord Dartmouth. Ο Λόρδος Ντάρτμουθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ερωτήσει για την Τουρκία. Είπατε στη γραπτή σας συνεισφορά ότι ανεξάρτητος και απαγγελματικός δικαστικός κλάδος είναι καθοριστική σημασίας για το κάτω δικαίου. Θεωρείτε ότι έχει τέτοιο ανεξάρτητο κλάδο η Τουρκία. Δεύτερον, στο πλαίσιο πάντοτε τη Τουρκία, να το θυμίσω και σε εσά και στου συναδέλφου, η στήριξη πρώτη προσχώρηση στην Τουρκία ήδη δίδεται. Ένα δι ευρώ ετησίω. Και παρόμοια ποσά έχουν προβλεφθεί μέχρι το 2020. Όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι όμω φυλακίζονται στην Τουρκία, περισσότεροι από ό,τι στο Ιράν και την Κίνα. Συμφωνείτε ότι όλη αυτή η στήριξη πρώτη προσχώρηση μήπω θα έπρεπε να ανασταλεί μέχρι να απελευθερωθούν οι δημοσιογράφοι. Και επίση μήπω συμφωνείτε μαζί μου ότι η στήριξη πρώτη προσχώρηση είναι ένα εργαλείο με το οποίο θα πρέπει να επιδιώξετε να επηρεάσετε την τουρκική κυβέρνηση. Ναι, όλα τα μέτρα αυτά βασίζονται στους ισχύοντες ε, κανόνες μας και κανονισμούς. Μόλις μια χώρα προσχώρησης ε, περάσει σε αυτή τη διαδικασία, πρώτης προσχώρησης, λαμβάνει χρηματοδότηση. Πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά εάν κάποιες εξελίξεις αντίκυνται τις αρχές αυτές, τη βασική μας την αντίληψη του ζητήματος, όμως κάποιες φορές τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από ό,τι φαίνεται. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το ζήτημα για να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Να επιτύχουμε αυτά που πολύ σωστά επικρίνατε είναι απαράδεκτο. Εντελώς απαράδεκτο ή οσδήποτε να φυλακίζεται. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την ελευθερία της έκφρασης. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Οπωσδήποτε θα το θέσω στις διαπραγματεύσεις μας και τις συζητήσεις μας με την Τουρκία προκειμένου να εξευρεθεί κάποια λύση. είναι κάτι που και μπορεί να διορθωθεί και δεν πρέπει να το αποδεχτούμε. Θα πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες αποκρίσεις. Όμω, με κάθε σεβασμό, κύριε υποψήφιε Επίτροπε, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να σα προσέξει ε, έστω και στο ελάχιστο η τουρκική κυβέρνηση, όπω δεν έχει κάνει και με του προκατόχου σα. σω ένα τρόπο πίεση είναι να προτείνουμε στι διαπραγματεύσει την αναστολή τη χρηματοδότηση πρώτη προσχώρηση. Και ο κύριο Γιούνκερ είπε καμιά προσχώρηση για την επόμενη πενταετία. Η δική μου εκλογική περιφέρεια δεν καταλαβαίνει γιατί 14 δις ευρώ έχουν προβλεφθεί για την ε, στήριξη πρώτη προσχώρηση όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια. Αυτέ οι χώρε τέλο πάντων. Ακριβώ. Γιατί η χώρα δεν θα λάβει 14 ε, δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ο συνολικό προπολογισμό ε, για τι χώρε τη διεύρυνση. Είναι, και μάλιστα είναι 11,7 δισεκατομμύρια, αν τα θυμάμαι σωστά. Και βεβαίως ε, πράγματι πρέπει να δούμε το ζήτημα αυτό. Πρέπει να το συζητήσουμε με τους ε, Τούρκους ομολόγους μας. Πράγματι δεν, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Εάν δεν είναι ικανοποιητικέ οι απαντήσεις, ε, πρέπει να δούμε πώς θα δράσουμε. Κύριος Επιτίδιος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο, όπως ανεφέρθη ήδη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, έχει δηλώσει ότι κατά την επομένη πενταετία δεν θα υπάρξει διεύρυνση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, οι συζητήσεις των υποψηφίων προς ε, ένταξη χωρών θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται. Μία από τις χώρες οι οποίες είναι η υποψηφία για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και η Φύρομ. Γνωρίζετε ότι η ενταξιακή διαδικασία της χώρας αυτής έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο λόγω της αντιδράσεως της ελληνικής κυβερνήσεως επειδή η κυβέρνηση της ΦΥΡΟΜ κατά παράβαση και των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Ελλάδα χρησιμοποιεί ως ε, επίσημο όνομά της το όνομα Μακεδονία που από την αρχαιότητα αποτελεί ε, ονομασία του μεγαλύτερου τμήματος της Βορείου Ελλάδος Πέραν όμως από το πρόβλημα αυτό, η Φύρομ δεν έχει, ε, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Κοπενχάγης. Θέλω να ρωτήσω ε, θα είναι η προσπά... πώς θα χειριστείτε, πώς χειριστείτε το, το ε, θέμα αυτό ώστε να υπάρξει ε, λύση που θα, που θα ε, εξυπηρετεί το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Listen to me. Your time is over. Συγχωρείτε, έχει τελειώσει ο χρόνος σας, Επίτροπε. Oh, Θεέ Παρακαλώ, έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Δεν ε, υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής επερώτησης. Ε, κύριε ε, Βουλευτά, η ΦΥΡΟΜ, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ε, συνδέεται με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για μένα τα προσεχή χρόνια γιατί βεβαίως δεν είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι η χώρα αυτή από το 2005 έχει το καθεστώς της υποψηφίας προς ένταξη χώρας, αλλά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και αυτό έχει μια αρνητική επίδραση στην ε, κατάσταση, ψυχική κατάσταση του πληθυσμού και επίσης για το λόγο αυτό επίσης ατόνισαν οι μεταρρυθμίσεις. Άρα λοιπόν συνολικά δεν πρόκειται για μια ικανοποιητική εξέλιξη και ως εκ τούτου ε, εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να βρεθεί τα προσεχή χρόνια μια λύση η οποία ασφαλώς δεν θα είναι εύκολη, έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος αλλά θα είναι αλλά είναι αναγκαία και αυτό προς όφελος του πληθυσμού και γι' αυτό θα ήθελα να υπάρξει εντολή να ξεκινήσουν, να δοθεί εντολή να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ε, ευχαριστώ που απαντήσατε και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί ο κύριος Πρόεδρος ήθελε να σε εμποδίσει να δώσετε αυτή την πολύ σωστή απάντηση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, η κυρία Βαλεντιάνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χάν, θα επιμείνω στην ε, πολιτική γειτονία προς τον Νότο, την Νότιο Μεσόγειο. Θυμάστε ότι από την Ευρακή από την Αραβική Άνοιξη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη και πιο έντιμη πολιτική όσον αφορά την ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεστε εκεί εσείς για να περάσετε από το επίπεδο των λόγων στο επίπεδο των πράξεων όσον αφορά την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως το σκηνικό εκεί είναι εξαιρετικά σύνθετο. κάθε χώρα συνιστά ένα κόσμο από μόνη της. Αλλά θεωρείτε ότι είναι ε, σωστό να εφαρμόζουμε την αρχή περισσότερο για περισσότερο όταν την εφαρμόζουμε στις, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, χρειάζεται ή προποθέτει μάλλον τη χάραξη μιας ιδέας στρατηγικής που εμπίπτει στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέεται με την ε, εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έλεγα εγώ, ε, εντάσσονται ή ανήκουν στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει το άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας που ορίζει επακριβώς το θέμα αυτό και θα πρέπει να εφαρμόζεται προς τα έξω και να λαμβάνεται υπόψη στις εξωτερικές μας δραστηριότητες. Θα ήθελα να απαντήσω συγκεκριμένα ε, στην ερώτησή σας ότι κυρίως η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών ε, αποτελεί ένα καθοριστικό μέτρο ούτως ώστε να ενισχύσουμε διαδοχικά, σταδιακά τα ανθρώπινα δικαιώματα της ελευθερίας, της ελευθερίας του λόγου, της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης. Και όλα αυτά ε, σε σύνδεση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι στο παρελθόν, σε αντίθεση με άλλους διεθνείς παράγοντες, ε, δεν ασχοληθήκαμε με θέματα των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, των social media, καθώς και τον ρόλο των, ε, της τηλεόρασης, για παράδειγμα. Ε, ε, θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τις δικές μας δυνατότητες για την εξασφάλιση θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων και την εγγύηση θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, σε αυτές τις κοινωνίες. Θα πρέπει λοιπόν να αθαρίσουμε τις απόψεις μας και θα πρέπει να σκεφτούμε νέες δυνατότητες επίλυσης. Ναι, όσον αφορά την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, γνωρίζετε ότι σε πολλές από αυτές τις ε, χώρες ε, περιορίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό το οποίο σας προτείνω, πέρα από τους προβληματισμούς, ε, να καταρτήσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τουλάχιστον αυτή θα ήταν η δική μου πρόταση. Να στηρίξουμε λοιπόν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που στις χώρες αυτής της λεγόμενης αραβικής άνοιξης βρίσκονται σε μια απελπιστική θέση. Ναι, ε, έχουμε, ε, ήδη, έχουμε σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού και αν ε, καταφέρουμε εδώ να ε, δούμε ποιοι είναι οι συνομιλητές μας, ε, θα βρεθεί αυτή η ευκαιρία, θα ανοίξει αυτός ο δρόμος. θεωρώ ότι παρόλα αυτά ήταν μεγάλη πρόοδος το γεγονός ότι όλες μας, σε όλες μας τις γειτονικέ χώρες οι φοιτητέ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέσχουν για παράδειγμα στο πρόγραμμα Erasmus Sin Άρα έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στην Ευρώπη και να σπουδάσουν εκεί και με τον τρόπο αυτό να εξοικειωθούν με τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή εμπειρία. Ε, ε, και ε, όχι βεβαίως για να φύγουν τα μυαλά αυτά από τη ε, χώρα τους. Θυμάστε τι είχε γίνει με εκείνο τον ε, ακαδημαϊκό, ο οποίος αυτό πυρπολήθηκε επειδή ήταν άνεργος. Αυτό που χρειάζονται λοιπόν οι άνθρωποι εκεί είναι να έχουν και μια προοπτική να εργαστούν εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ούτω ώστε άνθρωποι που έχουν μια ε, υψηλή μόρφωση και μια καλή κατάρτιση να μπορούν να μείνουν σε αυτές τις χώρες και να έχουν μια οικονομική προοπτική. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα και θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε συνολικά, σφαιρικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, υποψήφια Επίτροπε αντιμετωπίζουμε πρωτοφανείς απειλές ασφαλείας στη γειτονιά μας ε, και την Ανατολική και την Νότια. Τι άποψη έχετε για την ΚΕΠΑ και πιθανές αποστολές για να αποκαταστήσουμε την ειρήνη, την ε, ασφάλεια και τη σταθερότητα στην γειτονιά μας. Υπάρχει κάποιος ρόλος της πολιτικής διεύρυνσης ως κίνητρο για να διευκολύνουμε τον στόχο αυτό. Κοίταξτε, αυτό το ερώτημα μάλλον πρέπει να το θέσετε στην κυρία Μογκερίνη την επόμενη εβδομάδα. Βεβαίω για την πολιτική γειτονία οπωσδήποτε θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που υπάρχουν στην πολιτική γειτονία και οτιδήποτε σχετίζεται με τα ζητήματα ασφαλείας, αλλά είναι κάτι που πρέπει να αναπτύξουμε, αλλά δεν αποκλείω το να βρεθεί κάποιος κοινό τόπος και να υπάρχει μια αμοιβαία στήριξη κοινών μέσων επιπροσθέτως. How are you going θα διασφαλίσετε τις ε, συμφωνίες ε, με Γεωργία, Μολδαβία και λοιπές ε, και την ορθή εφαρμογή τους χωρίς ε, παρεμβολές. Ε, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Αλλά οπωσδήποτε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμόσουμε τις συμφωνίες που έχουμε με τους εταίρους μας. Αν δεν γίνουν τα πράγματα θα δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε. Αλλά ναι, επί της αρχής ε, είμαι αισιόδοξο. Είναι συμφωνίε ε, τι οποίες διαπραγματευόμασταν μήνες και χρόνια. Και βεβαίως ε, μέρος της διαδικασίας ήταν η ενημέρωση και η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία αμφιβολία για την ικανότητα εφαρμογής. Ε, ίσως εσείς σκέφτεστε κάποια πολιτική επιρροή, αλλά σας διαβεβαιώ πως η Ένωση θα είναι αυστηρή όσον αφορά την τήρηση των ε, συμφωνημένων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χάν, Θα επανέλθω στη συμφωνία με την Ουκρανία, ειδικά στις συνθήκες που οδήγησαν στην αναβολή της. Και έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πώς η Κομισιόν στο μέλλον θα ενημερώνει τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μέσω των ε, κανονικών διόδων και όχι να τα μαθαίνουμε από τον τύπο. Δεύτερον, μπορείτε να φροντίσετε και οι μελλοντικές ε, συμφωνίες ε, να λαμβάνουν υπόψη θεμελιώδη δικαιώματα, παραδείγματος χάρη οι πρωτομισιακές συμφωνίες για το εμπόριο. Και το αποτέλεσμα που είχαμε στην Ουκρανία νομίζω αποτελεί απόδειξη ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα στρατηγική σκέψη. Ποια διδάγματα αντλήσατε, ειδικά όσον αφορά και τις ε, συμφωνίες τερική σχέσης με την Νότια Μεσόγειο. Ναι. Για το πρώτο θέμα, κανείς δεν μπορεί να χαίρεται για το πώς ε, εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά από την άλλη, ε, σε γενικές γραμμές θα έλεγα πως είχαμε ένα μέτρο το οποίο λειτουργήσε ε, για να καταλήξουμε σε μια κατάπαυση του πυρός που επίσης στηρείται. Ε, δεν νομίζω να γίνει ρουτίνα το ζήτημα αυτό. Οπότε νομίζω μπορούμε να το θεωρήσουμε μια εξαιρετική ε, κατάσταση και η οποία βεβαίω απαιτεί εξαιρετικά μέτρα και οπωσδήποτε αυτά δεν προσφέρονται ε, για ιδανική αμοιβαία ενημέρωση. Ε, για το δεύτερο. Να σου πω την αλήθεια πρέπει να το δω και εγώ. Δεν έχω εξοικειωθεί με το θέμα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Η τρίτη ερώτηση ποια ήταν διδάγματα από τη στρατηγική κατάσταση. Ναι. Κοιτάξτε. Εγώ δεν βλέπω πλην της ε, αντιπαράθεσης ε, κάτι το οποίο ε, ήταν θα έλεγα ένα στρατηγικό λάθος. Ήταν μια διαδικασία που ε, κυλούσε επί σειρά ετών και τελικά νομίζω πως ε, η ενίσχυση και των ε, εμπορικών σχέσεων ε, νομίζω μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση και της ε, ελευθερίας και της δημοκρατίας στις χώρες με τις οποίες αναπτύσσουμε τέτοιες σχέσεις. Uh, Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, κατά πρώτον καλή τύχη στην τόσο δύσκολη δουλειά σας για τη γειτονία που θα πρέπει να περάσει από τον κύκλο πυρών σε ένα κύκλο φιλίας. Η ερώτησή μου είναι πόσο σημαντικό είναι για εσά και τι σκοπεύετε να κάνετε για την ενέργεια και την ανεξαρτησία μα από το φυσικό αέριο και γιατί μέσω τη συμφωνία σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Ουκρανία, Ένωσης-Ουκρανία-Σωστή η Ουκρανία να μπορεί να είναι ελεύθερη και χωρί εξωτερικέ πιέσει να μπορεί να επιλέξει πώ θα εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία. Δεύτερον, αυτή η ανεξαρτησία και πάλι από το φυσικό αέριο πως θα επιτρέψει στα κυρίαρχα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν ελεύθερες επιλογές ε, και χωρίς να υποκύπτουν στους εκδιασμούς της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, ήδη με την ε, τρέχουσα ιδιότητά μου ως Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής έχω προτείνει νέους κανονισμούς με συγκεκριμένα στοιχεία που στόχο έχουν να πετύχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανεξαρτησία της Ευρώπης από εξωτερικές πηγές ενέργειας να περιοριστεί. Αυτό ήταν μέρος των καθηκόντων μου και ήδη του χαρτοφυλακίου που είχα αναλάβει. Όμως, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι η ενέργεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ζήτηση για ενέργεια είναι πραγματικά ένα στοιχείο ευάλωτο γιατί ε, το ευάλωτο χαρακτήρα που μπορεί να δημιουργείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε διαφορετικούς πόρους για να προστατευτούμε ενεργειακά, αλλά και διαφορετικές μορφές ενέργειας. Αυτό μας καθοδηγεί στο να προβλέψουμε και νέες ε, γραμμές διανομής. Γι' αυτό έχουμε και το, ε, τον μηχανισμό Connecting Europe, διασύνδεση της Ευρώπης για καλύτερη διασύνδεση όχι μόνο εντός της Ένωσης, αλλά και προκειμένου να διασυνδεθούμε σωστά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η Ουκρανία επηρεάζεται κατά τον ίδιο τρόπο που μόλις εξήγησα. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε, να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να γίνει πιο ανεξάρτητη. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες βασικές προσπάθειες με την αντιστροφή των ροών. Όμως πρέπει να πω ότι και οι Ουκρανοί θα πρέπει να συνεισφέρουν στην όλη προσπάθεια. Η αγορά της ενέργειας στην Ουκρανία και επιτρέπει αλλά και θα χρειαζόταν κάπως μεγαλύτερη διαφάνεια και για τους Ευρωπαίους ε, φίλους τους. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε από όλες τις διαφορετικές σκοπιές το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ πρόεδρε Μπρόκ. Επίτροπε Χάν, δύο παρατηρήσεις και δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι η πείρα σας ως Επιτρόπου της Περιφερειακής Πολιτικής σας δίνει ε, τη δυνατότητα να εφαρμόσετε την αρχή της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης σε όλες τις χώρες και αυτών της διαδικασίας διεύρυνση και γειτονία. Έπειτα, εφόσον υπάρχουν σαφεί περιορισμοί για τι μελλοντικέ διευρύνσει, θα έχετε πολύ σαφέ καθήκον να ε, προβάλλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ω μοντέλο και ω παράδειγμα στι χώρε αυτέ που έχουν ε, ε, ενδεχομένω ευρωπαϊκή πορεία. Τώρα για τη Βοσνία και Ζεγοβίνη που δεν αναφέρατε στην εισαγωγική σα ομιλία, θα ήθελα να μου πείτε πώ βλέπετε τι εξελίξει μετά τι εκλογέ τη 12η Οκτωβρίου και πώς θα φροντίσετε ευάλωτα μέρη του πληθυσμού να έχουν πλήρη ε, εθνικά δικαιώματα, ειδικά στην Κροατία. Ε, για την αποκέντρωση των ορισμένων τμήματων του Γκάνσκ, τι θα γίνει με την ε, Ουκρανία και τα σύνορά της και την ενσωμάτωση αυτών των περιοχών. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας, διότι η αποκέντρωση σε κάθε περίπτωση είναι καλή και ελπιδοφόρα και συνήθως επιτυχής διαδικασία. Έχει να κάνει με την ανάληψη ευθυνών και την διαφύλαξη κάποιων αρχών. Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των ε, υπάρχουσων εντάσεων. Σε ό,τι αφορά τη Βοσνία και Ζεγοβίνη, μετά τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου, νομίζω υπόθηκε και σε μια από τις πρώτες μου απαντήσεις, θα καταβάλω προσπάθειες να έχω αμέσως επαφές με τους ίδιους τους βασικούς ηθήνοντες για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μέχρι τώρα είχαμε πολύ περιορισμένη πρόοδο όμως νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και να προσποθήσουμε να περάσουμε από τη λογική Dayton ίσως τη λογική των Βρυξελών περισσότερο. Να ξεπεράσουμε αυτό το τέλμα που υπάρχει στη χώρα και να μην αποδεχτούμε την κατάσταση ως έχει γιατί είναι όντως απαράδεκτη. Mr. very good afternoon. Το κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Η προηγούμενη Επιτροπή έθεσε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την δικαιοσύνη στην καρδιά της διαδικασίας διεύρυνσης. Εσείς προτίθεσα να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο. Και το δεύτερο εργαλείο για την πολιτική γειτονία ήταν, μας χαροποίησε που διαβάσαμε ότι ήδη έχετε δεσμευτεί στον στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφέρατε την ε, σύνδεση των, ε, της πολιτικής με την παροχή οικονομικής συνδρομής. Θεωρήσα, ε, θεωρείτε κύριε Επίτροπε ότι η έκβαση αυτής της συζήτησης τελικά θα καθορίσει την χάραξη προτεραιοτήτων εκ μέρους της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Βεβαίως είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η έκφαση των κοινών μας προβληματισμών θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις στην περιοχή αυτή. Ε, και πραγματικά μπορώ να βασιστώ στην εμπειρία που έχω ως επίτροπος επιφορτισμένος με την ε, περιφερειακή πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη. Ε, και θεωρώ ότι μία προτεραιότητά μας στο μέλλον θα έπρεπε να είναι να εργαστούμε επί τη βάση πολύ συγκεκριμένων προγραμμάτων τα οποία θα έχουν σαν σκοπό να συνδέσουν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων όχι μόνο μέσω λόγων αλλά μέσω έργων. Όταν μιλάμε λοιπόν για διασύνδεση της, ε, όσον αφορά τον ε, εφοδιασμό με ενέργεια ή τις ε, μεταφορές. Εάν τα επεξεργαστούμε αυτά με έναν ευφυή τρόπο, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα κονδύλια μας και θα δημιουργήσουμε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα χρήσιμα για τον ε, λαό των περιοχών αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Επίτροπε και από τη δική μου πλευρά σας εύχομαι το καλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι οι χώρες ε, ε, με ευρωπαϊκές ε, φιλοδοξίες, αν θέλετε, πρόσκειται στην Ευρώπη, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τις πρώην ε, κομμουνιστικές χώρες. Κύριε Επίτροπε, θα εργαστείτε στην ε, κατεύθυνση της συμβιλίωσης και αναφέρομαι εδώ στην περίπτωση της Σερβίας όσο και το άνοιγμα των αρχείων που περιλαμβάνουν στοιχεία σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούν ε, τμήμα της ε, πολιτισμικής μας ε, κληρονομιάς. Θα εμποδίσετε τους κομμουνιστές να αναλάβουν θέσεις κλειδί γιατί μέχρι στιγμής το ότι έγινε με το άνοιγμα των αρχείων της ΚΑΓΚΕΜΠΕ στη Μόσχα ήταν μια ψευδέστηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αναφερθήκατε στην ε, θέση του Κοινοβουλίου και βεβαίως θα το συμπεριλάβουμε στις διαπραγματεύσεις μας, αλλά και πάλι θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε ε, πάσης ε, φύσεως ε, επιλεκτική άσκηση δικαιοσύνης. Ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ίσο τρόπο όλους τους τέρους μας, όλα τα μέλη μας και βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ιστορικό παρελθόν από την άλλη και αυτό δικαιολογεί βεβαίως τα σχόλια και την πρότασή σας και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και να τα επεξεργαστούμε με ένα σωστό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάν. Ένα ερώτημα όσον αφορά τη Σερβία. Ο κύριος Φίλε ε, κατά την επίσκεψή του στο Βέλγιο έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες για τη χώρα. Πρώτον, οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, ε, κράτος δικαίου ε, και καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο μιας ευρείας μεταρρυθμίσης της δημόσιας διοίκησης. Και τρίτον, ε, ομαλοποίηση των σχέσεων με το Κόσοβο, με το Κωσυφοπαίδιο και συμφιλίωση στην ευρύτερη περιοχή. Συμμερίζεστε την άποψη του κυρίου Φίλε και πώς αξιολογείτε την, ε, τις μεταρρυθμίσεις στη Σερβία. Κοιτάξτε. Η Σερβία επέδειξε τους τελευταίους μήνες ε, πάρα πολύ καλή διάθεση και η νέα κυβέρνηση επίσης νομίζω είναι δεσμευμένη και στη διαδικασία αυτή. Ελπίζω, ελπίζουμε όλοι πως ε, όταν αποκτήσει καινούργια κυβέρνηση το κοσφοπέδιο θα επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις ε, σε πολιτικό επίπεδο. Σε τεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο υπαλλήλων ε, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Αλλά λόγω της έλλειψης ε, πολιτικής στήριξης η συμπερίληψη στο άρθρο 34 είναι, το, στο κεφάλαιο 34 είναι σημαντική και νομίζω αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα του γιατί χρειάζεται χρόνος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Γιατί όπως είπαμε το θέμα δεν είναι απλά να αλλάξει ένας νόμος ε, ή να συμφωνήσουμε κάτι αλλά να ε, επιδειχθεί πως υπάρχει συγκεκριμένη πρόοδος. Και ε, αυτό χρειάζεται χρόνο αλλά ειδικά για την Σερβία αυτή τη στιγμή είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Φαγιόν, ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Έχω μια-δυο ερωτήσεις σε σχέση με τη Σερβία. Αντιθέτως με άλλες υποψήφιες χώρες, η Σερβία ήταν η μόνη που δεν έλαβε μέτρα κατά της Ρωσίας πώς θα πείσετε τη χώρα αυτή και άλλους να ακολουθήσουν ε, την πορεία και τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περίπτωση και σε παρόμοιες περιπτώσεις. Μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική θα δραματίσετε καθοριστικό ρόλο για το διάλογο μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Έχετε κάποια συγκεκριμένη στατική για το Κωσυφοπέδιο και υπό το φως της τρέχουσας κρίσης ε, και την προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης. Πέντε είναι οι χώρες που ακόμη δεν αναγνωρίζουν το Κωσυφοπέδιο. Ε, εσείς πώς θα αναλάβετε διαμεσολαβητικό ρόλο στην Ποσνία ελζεγοβίνη αμέσως πριν τις εκλογές. Θα συνεργαστείτε με τα πολιτικά κόμματα για να υπάρξει εφαρμογή των συνταγματικών ε, αλλαγών που απαιτούνται ή θα ακολουθήσετε διαφορετική προσέγγιση. Ευχαριστώ. ότι η Σερβία εδώ έχει προσφέρει στην ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων και είναι μια απόδειξη για το γεγονός ότι κάποια πράγματα χρειάζονται χρόνο. Και επίσης είναι απόδειξη για το γεγονός ότι δεν μπορούμε μια νυχτή να καταλήξουμε σε, σταθερά, σε μόνιμα αποτελέσματα. Βεβαίως ε, η σερβική κυβέρνηση θα πρέπει να προβληματιστεί σχετικά γιατί εφόσον ενδιαφέρεται για την ένταξη ε, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις θετικές εκ μέρους των υποψηφίων χωρών. Και ε, κατά κανόνα διαπιστώνουμε ότι εναπόκειται στις ίδιες τις υποψήφιες χώρες να καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα, σε μια θετική έκβαση. Όσον αφορά το κοσυφοπαίδιο, εδώ έχει, υπάρχει μια δυναμική η οποία δεν πρόκειται να ανακοπεί από τις 15 χώρες που δεν αναγνώρισαν μέχρι στιγμή στο Κόσοβο. Νομίζω ότι εδώ έχουν αρχίσει να κινούνται τα πράγματα, αλλά και αυτό θα είναι αντικείμενο της εργασίας της, ε, υψηλής, της ΥΠΑ ε, εκπροσώπου και εγώ από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να κινήσω εδώ τα πράγματα, γιατί η κατάσταση που έχει δεν είναι ικανοποιητική. Και όσον αφορά την Βοσνία Ζεγοβίνη, ε, νομίζω ότι έχω κάνει ξεκάθαρο ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί η κατάσταση που επικρατεί εκεί με μηδενική πρόοδο εδώ και πολλά χρόνια ασφαλώς δεν είναι μια ευκταία κατάσταση και ελπίζω ότι μέσω της ένταξης της Κροατίας και της ε, δέσμευσης της Σερβίας και της ε, ιδέας μιας ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας ε, στον τομέα των συγκοινωνιών, των μεταφορών, της ενέργειας κλπ. Ε, σταδιακά και μέσω πραγματικών δεδομένων θα δημιουργηθεί μια κατάσταση τελικά de facto η οποία ε, θα έχει και μια θετική επίδραση στις πολιτικές εξελίξεις. Euh, κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, ε, ίσως ε, ε, έχουμε ξεχάσει την Νότια Ευρώπη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι επενδύσεις στην Νότια Ευρώπη εκ μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειωθεί κατά 20% και είχαν τα αρνητικά αποτελέσματα που γνωρίζουμε. Ε, στη συνέχεια της διαδικασίας της Λισαβόνας η Ένωση για τη Μεσόγειο το 2008 εκτροχιάστηκε. Εσείς προτίθεστε στο πλαίσιο της δικής σας θητείας να αναλάβετε μια πρωτοβουλία ούτως ώστε να μην αποκοπεί εντελώς η Ευρώπη από το Νότο ε, σήμερα οι πρώτοι επενδυτές στην Νότια Ευρώπη είναι οι χώρες BRIC, οι Κινέζοι. Και εμείς ε, τους έχουμε ε, κατ' ουσία εκχωρήσει το δικό μας ρόλο. Και νομίζω ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία. Εσείς προτίθεστε να φτιάξετε μια νέα ισορροπία και τι πρωτοβουλίες θέλετε να πάρετε για την Ευρωμεσόγειο που σήμερα πάσχει θα ήθελα να πω απευθυνόμενος προς την αίθουσα και εκτός της αιθούσης ε, ε, προς όσους ίσως έχουν την εντύπωση πως κοιτάμε μόνο ε, ανατολικά πως θα έχουμε όλα κατά νου είχαμε και το ερώτημα του κυρίου Πρέντα απάντησα πως κοιτάω και τα δύο δεν είναι μόνο ο Νότος, ούτε η Ανατολή. Είναι και τα δύο. Οτιδήποτε συμβαίνει στη γειτονιά μας έχει την αμέριστη προσοχή μας. Γιατί έχει άμεσες επιπτώσεις στην κατάστασή μας. Αν σκεφτούμε παραδείγματος χάρη τις ροές προσφύγων. Από την άλλη βλέπουμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες, ε, τις οικονομικές πρέπει να μας αποσχολήσει αυτό. Και βεβαίως είναι και στο άμεσο συμφέρον μας ε, να δούμε και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρεπούς ε, ζωής, ε, της αυτοδιάθεσης, αλλά, όπως είπα, πρέπει να έχουμε ως οδηγό το άμεσο ευρωπαϊκό συμφέρον. Και βεβαίως αυτό είναι από τον δακτύλιο αυτό της ε, φωτιάς να οδηγηθούμε σε έναν δακτύλιο ε, φίλων. Τέλος πάντων δεν είμαι τόσο αισιόδοξο, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να σβήσουμε κάποιες από τις φωτιές αυτές στη γειτονιά μας. Και εκεί πέρα νομίζω ακριβώς ε, η εταιρική σχέση με τις χώρες Μεσογείου είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο. Κύριε υποψήφοι ε, επιτροπέ, ερωτήσει μου αφορούν την Τουρκία. Το μπλοκάρισμα των ε, κεφαλαίων που οφείλεται και στη μη εφαρμογή του πρωτοκόλου της ε, Άγκυρας οδήγησε τον προκάτοχό σας, τον κύριο Φίλου, να ξεκινήσει τη λεγόμενη θετική ατζέντα. Εγώ θα ήθελα να δω πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα και πώς θα φέρετε την Τουρκία πιο κοντά στο να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει πλήρω το κεκτημένο. Είστε παραδείγματο χάρη υπέρ του να ξεκινήσουν να ανοίξουν νέα κεφάλαια για να εκμεταλλευτείτε πλήρω ε, την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωση που έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος, η οργανωτική δομή της Γενικής διεύθυνση Διεύρυνσης μια που η ομάδα εργασίας για τους Τουρκοκύπριους πήγε στην ε, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής. Πώς συνεισφέρει αυτό στην ε, ε, επιθυμητή επανένωση του νησιού. Για την πρώτη σας ερώτηση, νομίζω πως η προσέγγιση του Επιτρόπου Φίλε ήταν η σωστή και οπωσδήποτε δεν χαίρεται και δεν είναι ικανοποιημένο ε, με αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής. Αλλά οπωσδήποτε αυτή η προσέγγιση ήταν σωστή και ε, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Και, και το επαναλάβω, ε, οι τουρκικές αρχές πρέπει να μετακινηθούν, έχουμε συγκεκριμένους όρους, συγκεκριμένες συμφωνίες, υπάρχει το πρωτόκολλο της Άγκυρας και όσο δεν κληρώνονται αυτοί οι όροι, υπάρχουν εμπόδια ε, για να ανοίξουν νέα κεφάλαια. Αλλά μόλις συνάντησα τον νέο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ε, είχε μόλις παρουσιάσει ένα στρατηγικό έγγραφο για το πώς θα ξαναξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το αξιολογήσουμε αυτό αλλά όπως είπα είναι θέμα συγκεκριμένων πραγμάτων που πρέπει να κάνει η Τουρκία για να είναι αξιόπιστη και αυτό πρέπει να φανεί σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν για να βρούμε νέες ευκαιρίες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα κεφάλαια που δεν έχουν ανοίξει για τη νέα δομή τώρα. Αυτό είναι κάτι πρέπει να το δούμε. Νομίζω πως η μετακίνηση της ομάδας εργασίας στη Γενική Διευθύνση Περιφερειακής Πολιτικής οπωσδήποτε ε, έχει το σκεπτικό ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα έργα και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής έχει τις δυνατότητες, τη γνώση για να δει τη συγκεκριμένη εφαρμογή επιτόπου. Και πάλι Ε, είναι αυτή ίσως άλλη μια ευκαιρία στενότερης συνεργασίας ε, μεταξύ των δύο μερών ε, που μπορεί ελπίζουμε να οδηγήσει σε επανένωση του νησιού. Κύριε Χάν, ανησυχούμε ιδιαίτερως για την ευάλωτη κατάσταση που επικρατεί μετά την κρίση στη Λόρδα της Γάζας και την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση. Πρώτον, κάποια συγκεκριμένη δράση μπορείτε να σκεφτείτε για την μόχλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υπέρβαση των προβλημάτων με το Ισραήλ. Δεύτερον, πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστίνη πηγαίνει στους Παλαιστινίους πολίτες και τους ωφελεί. Ποια είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας. Και ε, τρίτον, ποια ε, άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου από, τον, ε, από την Κύπρο. Πολλές από τις ερωτήσεις σας θα έπρεπε να απευθύνονται στην κυρία Μογκερίνη. Δεν είναι ότι δεν θέλω να απαντήσω, αλλά πρέπει να είμαστε συντονισμένοι διότι έχουν πολιτικό χαρακτήρα αυτά τα ζητήματα και είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. εξ όσων καταλαβαίνω εγώ, θα πρέπει να εξυπηρετήσω τι δικέ τη προσπάθειε με τα εργαλεία και του μηχανισμού που διαθέτουμε στην πολιτική γειτονία, ώστε να μπορέσουμε από κοινού να βελτιώσουμε την κατάσταση και να συμβάλλουμε στην επίλυση, στην εξέβρεση λύσης. Σε ό,τι αφορά τον διάδρομο, νομίζω πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάνουν τα τρόφιμα και τα υπόλοιπα αγαθά στους πολίτες της ε, Γάζας είναι μέρος της διαδικασίας ειρήνευσης αυτό, όμως θα πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες και στη συγκεκριμένη περίπτωση ηγετικό ρόλο έχει η κυρία Μογκερίνη. Δεν αποποιούμε καμίας ευθύνης, όμως είναι ένα παράδειγμα, για να μην σας πω το πρώτο παράδειγμα, της αγαστής συνεργασίας που θα έχουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα βρίσκομαι. Η ελευθερία του τύπου ως προϋπόθεση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα καθώς η τέταρτη εξουσία είναι σημαντικό κομμάτι μιας δημοκρατίας και βλέπουμε ανησυχητικέ εξελίξεις ειδικά σε υποψήφιες χώρες, τα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία, ε, υποχωρεί η ελευθερία του τύπου και είπατε πως η ελευθερία έκφρασης ε, και πληροφόρηση τα ανεξάρτητα ΜΜΕ είναι για εσάς ε, βασική προϋπόθεση των διαπραγματεύσεων και Είπατε κάποια πράγματα, αλλά θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριμένο. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να μπει η ελευθερία του τύπου πιο ψηλά στις διαπραγματεύσεις δεδομένης της κατάστασης σε αυτές τις χώρες ε, και μάλιστα βραχυπρόθεσμα. Yeah. Νομίζω πως μάθαμε τα μαθήματά μας και ανοίξαμε τα σχετικά κεφάλαια πρώτα. Εκεί όπου μιλάμε για κράτος δικαίου, για ελευθερία γνώμης, για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ε, για διαφάνεια. Τα μάθαμε αυτά τα μαθήματα και χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο και στο Μαυροβούνιο και στην Σερβία ήδη και αυτά τα κεφάλαια θα είναι ταυτόχρονα και τα τελευταία που θα κλείσουν. Και βεβαίως ε, επανερχόμαστε συνεχώς στο ότι τα κεφάλαια αυτά ε, έχουν στόχο ε, πέρα από την ένταξη ή το κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να επιτύχουμε κάποιες άλλαγες, κάποια πρόοδο και εδώ πέρα πάλι επαφίεται στις ίδιες τις χώρες το πόσο γρήγορα θα ανταποκριθούν στις σαφές, σαφείς απαιτήσεις ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτό εξαρτάται τελικά το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν ε, βεβαίως δούμε τις φιλοδοξίες των χωρών αυτών και των λαών τους, νομίζω πως έχουν συμφέρον να ενταχθούν και νομίζω ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει στους λαούς τους είναι σημαντικό μέσο πίεση στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, εμείς ε, ε, πάντοτε διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε καλές ε, προθέσεις αλλά η Ρωσία εμποδίζει την περαιτέρω διεύρυνση. Πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Θα πρέπει να βάλουμε τις υποψήφιες χώρες πιο γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε μια απάντηση στη Ρωσία και θα αντισταθούμε στην πίεση που ασκεί η Ρωσία ή ε, γιατί αν δεν το κάνουμε η Ρωσία θα ασκήσει τις, ε, τους γείτονες χώρες υπό μεγαλύτερη πίεση δεύτερον, από την προηγούμενη εργασία σας στην Επιτροπή, πώς αντιμετωπίζετε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία One of Us. Νομίζω ότι καταρχήν είναι σημαντικό να δούμε ότι εναπόκειται στην κυριαρχία των ε, διαφόρων ε, λαών να αποφασίσουν, να κρίνουν ποιο δρόμο θέλουν να πάρουν και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, από τη δική μας πλευρά έχουμε κάποια συμφέροντα γιατί ενδεχομένω πρόκειται για υποψήφιες προς ένταξη χώρες ή για χώρες στην άμεση γειτονία μας και ανάλογα με το πώς ε, σχηματίζεται, πώς, υπάρχει, πώς δημιουργείται ο σχεδιασμός των δυνάμεων θα πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι το γεγονός ότι κάποιες υποψήφιες χώρες από μας έχουν ε, λάβει καθόλου αμεληταία ποσά προκειμένου να εξυγχρονίσουν τις κοινωνίες τους και να ενταχθούν στην Ευρώπη συνιστά σημαντικό πόλο έλξης έναντι μιας ε, κυρίαρχης ε, απόφασης που θα οδηγήσει τις χώρες αυτές προς την Ευρώπη. Και κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ερμηνεύσουμε τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για να υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές στο, στην προσπάθεια προσέγγισης της Ευρώπης προκειμένου να τις βοηθήσουμε να βελτιώσουν την κοινωνική τους κατάσταση και να αναπτύξουν υποδομές που θα καταστήσουν τις χώρες αυτές ε, πραγματικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών. Στο πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, ε, αν δούμε το 2007 στο 2013 είχαμε 12 δις ε, για τα μέτρα ενίσχυσης των χωρών αυτών για το 2014 έως το 20 ε, θα υπάρχουν 14 δις. Υπάρχει μια κοινωνική ποσόστοση πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια διασυνοριακή συνεργασία συγκεκριμένα. Θα οξύνετε τους ελέγχους ε, για, την, ε, τα κονδύλια όσον αφορά την δήλωση της Βαϊμάρης που υπογράφηκε τον Απρίλιο. Πώς θα εφαρμόσετε εσείς τα νέα, τις νέες ε, απαιτήσεις προτίθεστε να δημιουργήσετε θέσεις απασχόλησης, ε, θα εξασφαλίσετε ε, την ε, συνθήκες ασφάλειας για τις οικογένειες ή αποτελούν όλα αυτά τα στοιχεία τμήμα του πολιτικού σας οράματος. Κύριε Βουλευτά, ήδη σήμερα επισήμανα ότι όλες οι γειτονικές χώρες προς Νότο και Ανατολάς ε, θέλουμε στις χώρες αυτές ε, οι νέοι άνθρωποι να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εράσμους. Ε, και αυτό είναι ένα φιλικό μέτρο. Και βεβαίως προσπαθούμε να βελτιώσουμε και την οικονομική κατάσταση στις χώρες αυτές και αυτό για το δικό μας όφελος ούτως ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Αλλά θα ήταν αλαζονικό να ισχυριστούμε ότι η πολιτική μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Θα πρέπει μέσα των προγραμμάτων, σε πλαίσιο ή με την συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών να δημιουργήσουμε κάποιες πρωτοβουλίες ούτως ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα και να ενισχυθεί η οικονομία και με τον τρόπο αυτό να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες. Και αυτό με οδηγεί στο τελευταίο σημείο της ερώτησής σας, πράγματι ο έλεγχος των κονδυλίων ε, λαμβάνει χώρα και θα έχετε τη χαρά μια φορά το έτος, δεν ξέρω αν εσείς προσωπικά ή κάποιοι συνάδελφοι από την πολιτική σας ομάδα να ασχοληθούν με την ε, λεγόμενη απαλλαγή της Επιτροπής Χωρίς της Απαλλαγής και τα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολούνται μια φορά το χρόνο ε, ε, μάλλον ελέγχονται, γίνονται αντικείμενο ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο συντάσσει στη συνέχεια μια έκθεση ε, και αυτό περιλαμβάνει επίσης και τον ε, τομέα της ε, γειτονίας καθώς και της διεύρυνσης. Μέχρι τώρα η κατάσταση δεν ήταν πολύ ικανοποιητική, ωστόσο δείχνει ότι όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων, κατά κανόνα υπήρξαμε σωστοί. Και τελικά ο προγραμματισμός στις διάφορες χώρες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς διαμορφώνται τα αποτελέσματα του στρατηγικού διαλόγου και μετά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία στη δική σας εισφορά σχετικές προτάσεις για να δούμε πώς ε, θα γίνει ο αναπρογραμματισμός. Βεβαίως στην ε, περιφερειακή ε, πολιτική υπήρξε, ήταν πολύ σημαντικό το θέμα της αιρεσιμότητας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να επανέλθω στην Ουκρανία. Όπως γνωρίζετε η Ουκρανία λαμβάνει στήριξη τουλάχιστον 11 δις τουλάχιστον τόσα θα λάβει τα ερχόμενα χρόνια από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κινούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς και εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βεβαιωθεί ότι η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία ε, τη χάνει χρηστής διαχείρισης ε, βάσει των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης. Τι παρατηρήσεις μπορείτε να κάνετε σχετικά. Δεν έχω εγγύησει για το θέμα αυτό. Αλλά σας διαβεβαιώ. 11,7 δις για ένα-δυο χρόνια από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, Παγκόσμια Τράπεζα, ένα μείγμα διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης. Ο καθένας από αυτούς τους δωρητές έχει τους δικούς του μηχανισμούς παρακολούθησης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου για το πώς η συνεισφορά του δαπανήθηκε ακριβώς και πώς χρησιμοποιήθηκε. Το ίδιο και για τα κονδύλια που θα προέρχονται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και εδώ μηχανισμούς και εργαλεία, ώστε το ευρωπαϊκό χρήμα στην γειτονία και την πολιτική γειτονία να ε, δαπανάται και μάλλον να εκταμιεύεται απευθεία από τις αντιπροσωπείες μας, οι οποίες συνεργάζονται με οργανισμούς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτόπου. Έτσι λοιπόν κατευθύνονται τα κονδύλια μέσα από παγκόσμιους ενδεχομένου Παγκόσμιο κάποιες φορές φορεί με πολύ καλή στοχοθέτηση και πρώτο στόχο την ανοικοδόμηση της Ανατολικής Ουκρανίας. Αυτή είναι μια νέα πρόκληση και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανωθούμε. Αστρεβίτσιου, ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Χάν, με αυτό το διορισμό ε, σας ανατέθηκε μια ιστορική δουλειά και ιστορικές ευθύνες. Ποτέ προηγουμένω η γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν τόσο, ε, σε τόσο μεγάλη αναταραχή και δεν γνωρίζει τόσε πολλέ μεταπολέ. Ο προκάτοχός σα, ο κύριο Φίλε, κατάφερε την ανατολική γειτονία από μια ε, άλλη ιδέα να την εκφράσει σε χειροπιαστή πραγματικότητα με συγκεκριμένε συμφωνίε σύνδεση και συνεργασία. Εσεί, ε, κύριε Επίτροπε, εφόσον εγκριθεί ο διορισμό σα, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να πετύχετε, ποια είναι τα τρία στοιχεία που πιστεύετε ότι θα πρέπει να πετύχετε για να ονομαστεί επιτυχημένη η θητεία σα σε αυτήν την πεντέτεια. Και επίσης μια ακόμη ερώτηση για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Οι σχέσεις Δύση και Ρωσία είναι πολύ δύσκολε και ψυχρέ. Η, η ελίτ Ρωσίας έχει παραμείνει ε, εντό των τυχών του Κρεμλίνου τι θα κάνετε εσείς όμως για να απελευθερώσετε τον λαό της Ρωσίας και να εντείνετε τη συνεργασία με τους πολίτες της χώρας αυτής. Ευχαριστώ. Ε, πρώτον, για να προετοιμάσουμε τις περιοχές της διεύρυνσης και τις υποψήφιες χώρες, θα πρέπει να φροντίσουμε μόλις δούμε ότι κάποιοι έχουν την πρόθεση να προσχωρήσουν στην Ένωση, να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ήδη μια επιτυχία. αλλά για την ώρα δεν βλέπω να υπάρχει απέμπλοκη σε πολλές από τις ε, διαπραγματεύσεις που έχουν ε, βρεθεί σε τέλμα. Ε, ένα μικρό βήμα πρόοδου ίσως να ήταν κάτι τέτοιο, το να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Και το έχουμε ακούσει πριν από κάποιες δεκαετίες, ότι ένα μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα πολλές φορές. Ας δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις εκλογές στη Βοσνία Ριζεγοβίνη, με την πρώην κυκλοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κωσυφοπαίδιο ή την Τουρκία. Εκεί θα μπορούσαμε να περιμένουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Και για τη Ρωσία, για άλλη μια φορά, σημαντικό είναι να ε, διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Ακριβώς οι συνομιλίες μας να μην παύσουν και να δείξουμε στους Ρώσους φίλους και ομολόγους ότι η πολιτική γειτονίας, όπως είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως απειλή κατά της Ρωσίας. Θα είναι αμοιβαίως συμφέρον και για μας και για εκείνους να βελτιωθούν οι σχέσεις μας. Οι σχέσεις μας θα πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη και όχι τις αρνητικές εντυπώσεις, τον αρνητισμό. Πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Ο κύριος Νάρτ. Ε, κύριε Χάν, η Λέιδη ε, ε, μετά την, μετά την έρημο που άφησε η κυρία Άστον είναι πολλά υποσχόμενη η οάση που μας προτείνει ο κύριος Χάν. Ε, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία υπάρχουν πολλά κλειστά κεφάλαια. Αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι θεωρείται την Τουρκία πράγματι υποψήφια προς ένταξη χώρα και προτίθεται να στηρίξετε αυτή τη διαδικασία και να ανοίξετε κάποιο ε, κεφάλαιο. Δεύτερον, όσον αφορά το πάγμα τις σχέσεις με την Τουρκία. Δεν θεωρείτε ότι είναι ένας κίνδυνος να προσανατολιστεί η Τουρκία περισσότερο προς την Ασία, τη Μέση Ανατολή, ευθυγραμμιζόμενη ενδεχομένως και με τα ρωσικά συμφέροντα. Also, ich bin ein Είμαι πραγματιστής και πιστεύω ότι η Τουρκία για μας είναι ένας σημαντικός ε, εταίρος. Και για την Τουρκία εμείς ε, βεβαίως και είμαστε ο σημαντικότερος ε, εταίρος. υπάρχουν 120 δισεκατομμύρια ευρώ δικών μας επενδύσεων στην Τουρκία. Άρα λοιπόν η Τουρκία θα πρέπει να έχει ένα έντονο ενδιαφέρον, να έχει ε, πραγματικά ε, σωστές ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και λογικές σχέσεις και προσανατολισμένες προς το μέλλον. Εμείς από την άλλη έχουμε, ένα, έχουμε ορίσει ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο με ανοιχτό αποτέλεσμα όσον αφορά ε, μια μελλοντική προσχώρηση της Τουρκίας. Αυτή αυτά αποφάσισε το Συμβούλιο και αυτά θα πρέπει εγώ να τηρήσω το φίλο και θα παρακολουθήσω τις εξελίξεις αυτάς ως ε, πρώην Αυστριακός ε, Υπουργός θυμάμαι ε, τι γινόταν, ε, η Υπουργό Επιστήμης, ε, θυμάμαι ότι το κεφάλαιο το οποίο παρέμενε κλειστό ήταν το κεφάλαιο της επιστήμης. Είναι σημαντικό, όπως σας είπα, να συνεχίσουν οι συζητήσεις, αλλά βεβαίως όπως υπόθηκε εδώ κατά επανάληψη, ακριβώς εξασφάλιση των θεμελιδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός μιας κοινωνίας και συγκεκριμένα της τουρκικής, ε, θα πρέπει να είναι ε, ξεκάθαρος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όσον αφορά τον ρωσοτουρκικό άξονα δεν είπατε τίποτα. Ναι. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε για τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής στην επιστολή σας λέτε στον κύριο Γιόνκερ ότι χρειάζονται πολλές αποδείξεις για τους Ευρωπαίους πολίτες και σταθεροποίηση στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν είναι πολύ καλή η υπόσχεση αυτή όμω, διότι ο τίτλος χαρτοφυλακίου είναι διαπραγματεύσει για την προσχώρηση και την διεύθυνση. Αυτή τη στιγμή όμω το πρόβλημα και για δεν είναι τα πολιτικά μηνύματα. Δεν υπάρχουν διαφωνίε για την προσχώρηση των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που γεωγραφικά βρίσκονται στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο και έχουν σύνορα με πέντε, ε, κοινά σύνορα με πέντε κράτη-μέλη. Οι έξι αυτέ χώρε διασυνδέονται πολύ στενά μεταξύ του περισσότερο από ό,τι ποτέ στο παρελθόν με άλλε τι πιστεύετε λοιπόν για μια κοινή προσέγγιση και κάποιο είδους συντονισμένες προσπάθειες ώστε να υπάρξει μια διαδικασία προσχώρησης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. even though uh, Παρόλο που θα πρέπει ξεχωριστά να διαπραγματευτούμε και να συνομιλήσουμε με τις χώρες αυτές, τις χώρες αυτής της γεωγραφικής περιοχής. Και, αλλά βα, βασιζόμενος στις εμπειρίες μου ως Επιτρόπο Περιφερειακής Πολιτικής, πρέπει να πω το εξή. Είδαμε τι γίνεται με τις στρατηγικές για τις μακροπεριοχές, όπως ονομάστηκαν, τη στρατηγική του Δούναβη λόγου χάρη, ή την στρατηγική για την Αδριατική που οδεύει προς ολοκλήρωση. Εκεί κάποιες από τις χώρες, για να μην πω όλες, υποψήφιες ή ενδυνάμει υποψήφιες, συμμετέχουν πλήρως. Ένας από τους δικούς μου στόχους λοιπόν νομίζω θα είναι να βελτιωθεί η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο με τις χώρες αυτές αλλά και εντός της ίδιας της περιοχής. Τα σύνορα δεν σταματούν εκεί που τελειώνει η επικράτεια των κρατών μελών αλλά κάποιες φορές στην Κροατία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα υπάρχουν προεκτάσεις. Ε, εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ολόκληρης της γεωγραφικής αυτής περιοχής. Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε να συμβάλλουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Σακοράφα. Κύριε Χάνς, η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκληση στον εκδημοκρατισμό και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα συμμετείχε έμεσα ή άμεσα σε όλες τις επεμβάσεις στη λεκάνη της Μεσογείου. Αποτέλεσμα να έχουμε διάλυση κρατών, χιλιάδες αμάχους νεκρούς και εκτοπισμένοι σε Ιράκ, Συρία, Λίβανο, έξαρση φονταμενταλισμού, προέλαση Ισλαμικού κράτους, κατοχή και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Παλαιστίνη και Μαρόκο. Η Μεσόγειος έγινε ένα απέροντο υγρό νεκροταφείο αθώων. Επιπλέον, η Ένωση συνάπτει συμφωνίε σύνδεση και σχέσει με κράτη κατοχή που αδιαφορούν για τι αρχέ και τι αξίε τη, περιφρονούν το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο και αγνοούν επιλεκτικά διεθνεί συμφωνίε και αποφάσει. Συγκεκριμένα λοιπόν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και συνεργασία με την κυρία Μοργκερίνη. Τι πρωτοβουλίες θα πάρετε, πώς θα αναγκάσετε κράτη κατοχής όπως το Ισραήλ και το Μαρόκο να συμμορφωθούν, πώς θα αναγκάσετε το Ισραήλ να σεβαστεί τις διεθνείς αποφάσεις για τους επικισμούς, εξετάζετε το ενδεχόμενο χρήση του άρθρου 2 των συμφωνιών σύνδεσης για πάγωμά τους όσο παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι ή όχι. Σας ευχαριστώ. Uh, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του Μαρόκου φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην περίπτωση της Δυτικής Σαχάρας ε, και την πολιτική του επικισμού έχει ξεκάθαρη θέση ε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα για την Δυτική Σαχάρα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει σαφής εντολή του ΟΗΕ και από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς ε, στηρίζουμε και παρακολουθούμε αυτές τις ε, προσπάθειες αλλά δεν έχει και πολύ νόημα γιατί ξέρετε όπου λαλούν πολύ κοκόροι αργεί να ξημερώσει ο καθένας καλύτερα να κάνει αυτό που Πρέπει εμείς παρακολουθούμε πράγματι την εφαρμογή και όταν απαιτείται η δικιά μας ε, συνεισφορά, οπωσδήποτε θα συνεισφέρουμε. Κύριε Επίτροπε, σας χαιρετώ. Υποθέτω ξέρετε ότι εσείς και εγώ και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούμε να ταξιδέψουμε σε όλα τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εγκληματίες δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Εν τούτης υπάρχει μια περιοχή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Γιούγκερ, ούτε εγώ μπορούμε να επισκεφθούμε. Σας το απαγορεύει ο τουρκικός στρατός και αναφέρομαι στην πόλη της Αμοχώστου. Θέλω να μου πείτε αν θα επιχειρήσετε να επισκεφθείτε αυτή την πόλη, όχι απλώς γιατί είναι μια κίνηση σωστή, αλλά γιατί θα δώσετε μια τεράστια όθηση στο να παραδοθεί η πόλη στους κατοίκους της, αλλά και ίσως να επιληθεί το κυπριακό πρόβλημα. Θέλω να ξέρω λοιπόν αν θα επιχειρήσετε να κάνετε αυτό το βήμα, γιατί θα είναι προς όφελος όλης της Ευρώπης, θα είναι προς όφελος της Τουρκίας, γιατί στο τέλος τέλος εάν κινηθούν τα πράγματα στην επίλυση θα ανοίξει ο δρόμος και για την ίδια και θα πάψουν κράτη να κρύβονται πίσω από το Κυπριακό εμποδίζοντας την ένταξή της. Ευχαριστώ. Ναι, με την τελευταία, πρώτη-τελευταία πρότασή σας πράγματι τονίσατε κάποια πράγματα και κάποιες συμπεριφορέ που οδηγούν στο μπλοκάρισμα των συνομιλιών. Τώρα συγκεκριμένα για την αμόχωστο, εγώ είμαι νέος στην ε, διπλωματία θα ήθελα να έχουμε κάποια αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε θα μιλήσουμε με τους ειδικού. Καμιά φορά πρέπει να αναζητούμε και νέους δρόμους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω τίποτα συγκεκριμένο, αλλά οπωσδήποτε σημειώνω αυτό το οποίο είπατε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χάν, σας ευχαριστώ για αυτό το οποίο δηλώσατε ξεκάθαρα για την ανάγκη θεμελιωδών αλλαγών στην ε, πολιτική γειτονία και μιλήσατε για ε, όρους και για το ότι θα πρέπει από κοινού να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι χώρες και οι, ευρωπαϊκές και οι χώρες Η σύνοδος του Βίλνιους όμως έδειξε πως οι χώρες αυτές καθοδηγούνται σε ε, αντιπαλότητα με την Ρωσία. Και μάλιστα υπάρχει αυτό το δίλημα Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ρωσική Ομοσπονδία το οποίο είναι υψηλού πολιτικού κινδύνου για όλους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε συγκρόσεις ε, εντός ε, των κοινωνιών. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε για να μειωθούν οι συγκρούσεις και ειδικά με βάση την αυτοδέσμευση που αναφέρατε για την εξορόψη των συμφερόντων και θα πάτε ε, στο Κισνόβιο και στο Κίεβο δεδομένης δε και της ε, δέσμευσης που υπάρχει ε, για να γίνουν κάποιες χώρες κάτι μέλη. Κοιτάξτε. Οπωσδήποτε θα επισκεφθώ το στομότερο δυνατόν όλες τις χώρες ε, που είναι αρμοδιότητά μου. Και η Μολδαβία οπωσδήποτε είναι μια χώρα την οποία θα επισκεφθώ κατά προτεραιότητα. Έχουν εκλογές το Νοέμβριο. Είναι Βεβαίω θέμα της ε, κάθε χώρας το πώς θέλει να τοποθετηθεί στο μέλλον, τι ε, πώς θα διαμορφώσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διάφορες ε, δυνατότητες, ε, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί κάποια επεκτατική πορεία ή κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε λογικές σχέσεις με τους γείτονές μας. Όποιος θέλει να προσεγγίσει πιο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τον στηρίξουμε αλλά παραμένει κυρίαρχο δικαίωμα της κάθε χώρας και του λαού της λογικά να αποφασίσει. Είναι νομίζω σημαντικό και ελπίζω και από τη ρωσική πλευρά να βλέπουν έτσι τα πράγματα. Δεν ε, δεν τίθεται ζήτημα κάποια αντιπαράθεσης. Νομίζω είναι και προς το ρωσικό συμφέρον να επικρατήσει σε αυτές τις περιοχές ε, ευημερία, ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατικά συστήματα, τα οποία τελικά είναι και η βάση νομίζω του να μπορούν οι άνθρωποι να επιτύχουν περισσότερα και να έχουν περισσότερη ευημερία. Αυτή την πολιτική ακολουθούμε Αυτά τα μηνύματα θα ήθελα να στείλω. Και ελπίζω τελικά να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε χωρίς κυρώσεις. Αλλά, εάν ε, είναι αναγκαίο, δεν θα διστάσουμε. Γιατί οπωσδήποτε παραβιάσεις εδαφικής ακαιρεότητας ε, δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές και ελπίζω να καταλήξουμε ξανά σε ένα επίπεδο συζήτησης όπου θα μπορούμε να ζούμε και να έχουμε κάποια εξέλιξη χωρίς κυρώσεις. Η κυρία Κύριε Πίτροπε, η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία αυτή τη στιγμή ε, δεν μας αφήνει πολλές ελπίδες, αλλά υπάρχουν πολλές ανησυχίες ότι εσείς ως Επίτροπος ε, Γειτονίας ενδεχομένως ε, στην περιοχή αυτή θα έρθετε αντιμέτωπος με, ένα λεγόμενο, με μια λεγόμενη παγωμένη σύγκρουση όπως αυτή που γνωρίζουμε από την Απχαζία και την Υπερδνηστερία. Ποια είναι η δική σας στάση εδώ, ε, πώς θα πρέπει να το χειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα αποθετήσετε ε, ε, για τη, έναντι της των κυρώσεων και ποιες είναι οι προϋποθέσεις πλαίσιο που θα ισχύσουν στην περίπτωση αυτή. Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά την πάταξη της διαφθοράς και το κράτος δικαίου στην Ουκρανία. Αυτή ήταν η ισχυρότερη επιθυμία παράλληλα ε, με την ελευθερία και τη δημοκρατία στην ε, εξέγερση στην πλατεία Μαϊντάν. Ε, και πώς μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε θετικά εδώ. Απάντηση. Όσον αφορά την Ανατολική Ουκρανία, τα πράγματα εδώ είναι αρκετά ξεκάθαρα. Θα πρέπει να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ε, εδώ έχουν γίνει διάφορες προτάσεις και από τον, κύριο, από τον πρόεδρο ε, κύριο Ποροσέγκο ε, υπάρχει ο, ο, κύκλος, ο γύρος του, Ρουντ, του Μίνσκ συγγνώμη, και ελπίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο που βεβαίως είναι αρκετά επισφαλής γιατί η κατάπαυση πυρός παραβιάζεται συνεχώς. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξο ότι η εισαγωγή αυτού του διαδρόμου των 30 χιλιόμετρων ε, θα συμβάλλει στην διατήρηση της ειρήνης ενδεχομένως. Αλλά για μας ως Ευρωπαίους εδώ δεν υπάρχει καμία ενδιάμεση λύση όσο δεν έχει αποκατασταθεί η εδαφική ε, κυριαρχία και ακαιρεότητα. Ε, δεν μπορούμε να ενδώσουμε όσο δεν αποκατασταθεί η εδαφική ακαιρεότητα, δεν μπορούμε να ενδώσουμε στην Ρωσία. Όσον αφορά το άλλο θέμα, πιστεύω ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες του Ποροσέγκο να έρθει, να έρθει πιο κοντά η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινήσει μια προενταξιακή διαδικασία και κάτω από αυτό το πρίσμα να γίνουν και οι μεταρρυθμίσεις εκεί. Αναφέρθηκε σε 50-60 αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και θεωρώ ότι κάτι θα πρέπει να εννοεί με αυτές, όχι απλώς να αναφέρει έναν αριθμό. Ε, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να ασκήσουμε πίεση εφόσον αν θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά τους λαούς των γειτονικών χωρών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να έχουμε πιο στενές σχέσεις με αυτές τις χώρες, θα πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα και αυτά πηγαίνουν ε, στην κατεύθυνση των ετοιμάτων των εξεγερμένων στην ε, πλατεία Μαϊντάν, δηλαδή ε, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, διαφάνεια και δημοκρατισμός, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, και εγώ θα συνδεθώ με το ερώτημα του κυρίου Ράντο για την διεύρυνση. Ε, στην επιστολή σας λέτε, όπως είπε και ο κύριος Γιούγκερ, ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω διευρύνσεις τα προσεχή πέντε χρόνια. Και γιατί θα πρέπει οι πολίτες μας να χωνέψουν την ε, ένταξη 15 νέων χωρών. Για μένα αυτό ακούγεται κάπως ε, περίεργα, σαν να σηματοδοτεί το πέρας την, ε, της πολιτικής διεύρυνσης. Πώς θέλετε να εξασφαλίσετε οι Ευρωπαίοι πολίτες τα επόμενα πέντε χρόνια να χωνέψουν αυτή τη διαδικασία των προηγούμενων ετών κατά τρόπο που να συνεχίσει η διαδικασία διεύρυνση η οποία αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα του ειρηνευτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Νομίζω ότι θα πρέπει να... Α, η ερώτηση ήταν για την, διεύρυνση, για την προσχώρηση της Ισλανδίας. Εφόσον έχει φτάσει στο σημείο αυτό, έχει το κοινωνικό εκτιμένο, πώς θα αντιδράσετε, είχε ρωτήσει η κυρία Λούνατσεκ. Η απάντηση είναι ότι αν φτάσουν στο σημείο αυτό οι Ισλανδοί, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε γιατί εάν δούμε τι γίνεται με τους Αλής για παράδειγμα υπάρχει ένα περιθώριο συζητήσεων για το τι γίνεται στην Ισλανδία. Ε, και θα ήθελα να σας πω κάτι όπου εμείς οι Ευρωπαίοι πραγματικά θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Και το λέω σε κάποιος που έχει ασχοληθεί με το χώρο της οικονομίας εδώ και πολλά χρόνια. Εάν ε, ένας επιχειρηματικός όμιλος ε, είχε αναπτυχθεί ε, όπως έχει αναπτυχθεί η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, θα ανέμενε κανείς τελικά να ακολουθήσει φθήνουσα... δεν θα ανέμενε κανείς να ακολουθήσει φθήνουσα πορεία. βρισκόμαστε στην Ευρώπη των 28 Εάν το είχα μεταφέρει αυτό σε οικονομικούς όρους, θα μπορούσα να κάνω ως ασφαλή πρόβλεψη ότι θα ακολουθήσει χρεοκοπία. Ε, και εμείς ε, πραγματικά ε, καταφέραμε να μην επέλθει η χρεοκοπία ή τα καταφέραμε ε, βεβαίως να υπάρξουν ορισμένοι κλειδονισμοί αλλά να μην ε, χρεοκοπήσουμε ως Ευρώπη. Το οικοδόμημα στέκεται ακόμα στα πόδια του. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε υπερήφανοι και να έχουμε επίγνωση ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην κατάσταση που να είμαστε σε θέση να δεχθούμε την ε, επόμενη ε, διεύρυνση. Και ε, θεωρώ ότι βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια θετική προετοιμασία στις χώρες μέλη και αυτό το λέω σε επίτροπος διεύρυνσης να υπάρξει μια θετική προετοιμασία για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται μελλοντικά να αυξηθεί, να διευρυνθεί δηλαδή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Κάτι από τα οποία συμφωνούμε σε όλοι είναι ότι για τα οποία συμφωνούμε όλοι είναι ότι για την ήπια δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά τα πάει, αλλά για τον ρόλο που μπορεί να παίξει για την προστασία των, της κοινωνίας των πολιτών ε, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ακόμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως στην επιστολή σας μεταξύ των δεσμεύσεών σας ε, λέτε πράγματα που είναι πολύ καλοδεχούμενα. Όμως τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε ε, για τις χώρες της γειτονίας που δεν φαίνεται να στηρίζουν την κοινωνία των πολιτών τους, μάλιστα την ε, καταστρέφουν όπως την Αίγυπτο και αλλού. Εκεί τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει και θα μπορούσατε να είσαστε λίγο πιο ηχηρός όταν εκφράζετε τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ε, τάσεστε υπέρ της προστασίας των ε, οργανισμών που προστατεύουν την κοινωνία των πολιτών. Προς τον Νότο, θα πρέπει προσωπικώς να κοιτάξω, να βολιδοσκοπήσω τα πράγματα και να μετρήσω τις δυνατότητες και τις μέρημνες της κοινωνίας των πολιτών εκεί. Ε, στην Αίγυπτο υπάρχει και σχετικός νόμος που εγκρίθηκε πρόσφατα. Θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει λοιπόν. Καλά λέτε ότι πρέπει να είμαι πολύ χειρό στην έκφραση της φωνής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό ακριβώς και θα κάνω, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει κοινωνία των πολιτών και να προστατεύονται έτσι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εάν έχουμε μια πολυφωνική, πολύχρωμη κοινωνία των πολιτών, μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε στη δημοκρατία. Είναι προϋπόθεση για το δημοκρατικό πολίτευμα να υπάρχει ευρεία διαφοροποιημένη και ποικίλη κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει κονδύλια για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Όμως πρέπει να βεβαιωθούμε και να επαναποτιμήσουμε αν αυτά λειτουργούν αποτελεσματικά. Πού μπορεί να επέλθουν βελτιώσεις και τι γίνεται με την εκταμείευση και την δαπάνη κονδυλίων από την κοινωνία των πολιτών, γιατί ακριβώ θέλουμε βιώσιμα αποτελέσματα και πρόοδο. Νομίζω αυτό μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που μου ζήτησε ο κύριος Γιούνκερ να προτείνω, μία νέα αναδιαρθρωμένη πολιτική κοινωνίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά την Ουκρανία. Εσείς προσωπικά είστε υπέρ του να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα μας πείτε ότι δεν το έχετε σκεφτεί και άρα δεν έχετε συγκεκριμένη απάντηση. Εγώ θα έλεγα πως οι ακροάσεις αυτές έχουν στόχο να ακούσουμε την δική σας άποψη πέραν από την άποψη Κομισιόν. Ε, από τις ε, προηγούμενες ε, απαντήσεις σας έχουν εντύπωση πως λυπάστε για την καθυστέρηση της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Ισχύει αυτό ή όχι. Και τέλος, στην προπροηγούμενη απάντηση για τις περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέχεστε πως οι πλούσιες χώρες δεν θέλουν να ενταχθούν π.χ. η Νορβηγία και η Ελβετία. Και αυτές που θέλουν να ενταχθούν είναι πολύ φτωχές που θα αποτελέσουν βάρος οικονομικό στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Δέχεστε κάτι από αυτά. Δεν ξέρω, ναι, ίσως να αλλάξουμε και να καθίσω εγώ στο Προεδρείο. Λοιπόν, για την Ουκρανία. Ναι, είμαι και εδώ ρεαλιστής. Κάποιοι από μας είχαν πάει εκεί επί τόπου στο Μαϊντάν. Υπάρχει ενδιαφέρον επιθυμία της πλειοψηφίας των Ουκρανών όπως φάνηκε και στις τελευταίες εκλογές να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το στηρίξουμε νομίζω. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα τίποτα περισσότερο. Και πάλι νομίζω είχαμε μια αρεαλιστική προσέγγιση του Προεδρού Ποροσέγκο που έλεγε πως ε, ακόμα και η αίτηση ένταξης απαιτεί πολλές ε, μεταρρυθμίσεις και πρότεινε τα επόμενα 5-6 χρόνια να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα αποτελούσαν ίσως τη βάση μιας αίτησης, αλλά νομίζω πως απέχουμε ακόμα πολύ. Όχι μόνο χρονικά, αλλά και επί της ουσίας. Και από την άλλη Υπάρχει μια σαφής επιθυμία του Ουκρανικού λαού να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να την απορρίπτουμε. Τώρα. Για την διακοπή αυτή ε, κανείς δεν ε, ικανοποιήθηκε αλλά ήταν θα έλεγα ένα μέτρο που βοήθησε στην κατάβαση του πυρός. Και νομίζω πως όλοι θέλουμε να αποφύγουμε τα περαιτέρω θύματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως θύμισαν και άλλοι, η κρίση της Ουκρανίας έχει απομακρύνει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ανατολική γειτονία. Και ενώ οι πολίτες ασχολούν, ε, ανησυχούν για την Ρωσία, έχουμε ξεχάσει την γειτονία μας προς τον Νότο με την Αραβική Άνοιξη και όλες αυτές τις ελπίδε που τελικά εξατμίστηκαν με τις εξελίξεις της χώρας αυτές. Ετοιμάζεται λοιπόν μια ε, μεγάλη κρίση λόγω τη Λιβύη που ετοιμάζεται να γίνει ένα πραγματικά αποτυχημένο κράτος. Πώς θα μπορούσαμε εδώ να παρέμβουμε με την πολιτική γειτονία και πέραν των ε, συγκεκριμένων ε, ε, επιγουσών αναγκών πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια προληπτική δράση που είναι και αποτελεσματική. Βεβαίω η κρίση προς Ανατολά είναι πολύ σοβαρή, Όμω, με τόσε χιλιάδε μετανάστε να έχουν φτάσει στι ακτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 2014, είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε και με το τι γίνεται με την κρίση προ τον Νότο. Πώ μπορούμε λοιπόν να βρούμε τη σωστή ε, ισορροπία για την πολιτική γειτονία, ακόμη και γεωγραφικά, και πώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια προληπτική δράση ώστε να μην βρίσκεται κάθε φορά λύσει κομμένε και γραμμένε στι ανάγκε τη στιγμή, αλλά πιο μακροπρόθεσμε. Θέλω να σας ε, διαβεβαιώσω ότι ενδιαφερόμαστε και για το Νότο και όχι ε, επειδή η Αραβική Άνοιξη ήταν την Άνοιξη και τώρα είμαστε στο φθινόπορο, έχουμε πάψει να ενδιαφερόμαστε. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό στη γενική μας ε, διεύθυνση. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνο για το γεγονός ότι η κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή στρέφεται περισσότερο ε, προς ε, Ανατολάς. Εγώ θεωρώ ότι στη δική μας διεύθυνση δίνουμε και στις δύο περιοχές ε, την ίδια σημασία ε, και όσον αφορά την κατανομή κονδυλίων έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει και το προσωπικό. Με όλες τις σχολίες λοιπόν που υπάρχουν στον Νότο που δεν θέλω να τις αγνοήσω, γιατί βεβαίως υπάρχουν και θετικά παραδείγματα, αν δούμε για παράδειγμα τις εξελίξεις στην ε, την Ισία ή και την πρόοδο στο Μαρόκο ή στην Ιορδανία. Ε, βεβαίως δεν, είμαστε, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που επιθυμούμε, αλλά θεωρούμε ότι είναι δυνατό να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα εφόσον βεβαίως επιμείνουμε αρκετά. Υπάρχουν βέβαια άλλες περιοχές όπως η Λιβύη όπου απέχουμε τρομακτικά από το ευκταίο αποτέλεσμα και θα πρέπει να σπάσουμε το κεφάλι μας για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά την Επιτροπή και εμένα τον ίδιο δίδουμε αρκετή προσοχή προς ε, το νότο. Godātais κύριε Επίτροπε, ε, η επιβολή κυρώσεων έχει διαφορετικά αποτελέσματα ε, στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ίσως η έκφραση αλληλεγγύης θα ήταν πιο χρήσιμη. Εάν δούμε το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχετε αναλάβει, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πρόκειται να πάρετε κάποια μέτρα για να αποφύγετε αρνητικά για να έχετε αρνητικές, για να επιβάλλετε κάποιες οικονομικές κυρώσεις ε, στο νότο της Ευρώπης. Αλλά τι θα γίνει με τα οικονομικά προβλήματα. das ist, ε, Δεν είναι ε, η άμεση αρμοδιότητά μου, αλλά συζητήσαμε με τους συναδέλφους αυτό το θέμα για παράδειγμα με τις ε, ενισχύσεις στη γεωργία. Εγώ θεωρώ ότι αν ε, εδώ ε, υπάρχουν τέτοιες δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αλλά με αυτό θα πρέπει να ασχοληθεί το σύνολο της Επιτροπής και βεβαίως και οι χώρες μέλη που θα πρέπει να που θα ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτά. Ακούσαμε για αεροδρόμια. Εδώ ακούσαμε ότι κλείνουν αεροδρόμια και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Ουκρανία. Πόσα ε, χρόνια θα μας πάρει να αποφασίσουμε αν η χώρα θα παραμείνει ενωμένη, αν θα κατακαιρματιστεί ή αν θα ε, διαιρεθεί. Πόσο καιρό μπορούμε επίσης αυτούς που μας χτυπάνε στην πόρτα κατά αυτόν τον τρόπο να τους ε, ταπεινώνουμε. Τι θα γίνει με τη Ρωσία επίσης η οποία μας ε, υποβιβάζει διαρκώς και μας χλεβάζει. Επίσης τι θα γίνει με τον ε, Λουκασέγκο και την ε, δημοκρατία στη Λευκορωσία. Ξέρετε ότι 70% των Λευκορώσων που είναι πολύ κοντά στην Μόσχα θα ψηφίσουν την ε, προσχώρησή τους στην Ρωσική Ομοσπονδία και θα έχουμε το ρωσικό στρατό πολύ κοντά στα σύνορά μας. Ε, Κοιτάξτε. Συμπολίτική. ε, δεν έχω μάθει να ασχολούμαι με υποθέσεις αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και ε, προσπάθω πάντα να συνομιλώ με τη θεωρίας του μισογεμάτου ποτηριού και πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα και να μην δημιουργούμε καινούρια. Αυτό νομίζω πρέπει να μας ε, καθοδηγεί και ειλικρινά να σας πω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, νομίζω αρκετά υψηλό ηθικό ανάστημα, δεν χρειάζεται να κρύβεται και στη τελική ανάλυση άλλοι θα καταστούν. Καταγέλαστε και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να μας δώσετε μία συγκεκριμένη απάντηση για το εάν και πότε η Γεωργία θα κάνει κάποια βήματα προσέγγισης. Για, το λέω αυτό γιατί η Λετωνία την οποία εκπροσωπώ είχε μια παρόμοια εμπειρία. γιατί αυτό προσφέρει βεβαίως και κίνητρα στην χώρα. Εγώ είχα πάει στη Γεωργία, συναντήθηκα με τον πρόεδρο, την αντιπολίτευση και είναι ξεκάθαρη η επιθυμία τους να έχουν τουλάχιστον μία απάντηση όσον αφορά τις προοπτικές τους. Αν και ίσως είναι κάπως μακριά μία τέτοια προσωπική. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε εξ ονόματος Κομισιόν, πείτε μας την προσωπική σας άποψη. Ναι, ε, δεν μπορώ Όμω έτσι να αποδεσμευτώ τελείω και δεν το θέλω. Ο λαός της Γεωργίας ε, ξέφρασε την θέλησή του. Έχουμε κάποιες συμφωνίες, αλλά αν πάτε εκεί θα διαπιστώσετε πως πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα, ε, ανεξάρτητη δικαιοσύνη κτλ. Έχουμε κάποια θέματα. Και οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει μια διασφάλιση δίκαιης, ισότιμης ε, μεταχείρισης ε, και να μειωθούν οι κοινωνικές εντάσεις γιατί οπωσδήποτε ε, υπάρχει εδώ πέρα αν θέλετε μια Υπάρχει ένας ρυθμός ε, και μια δυναμική που έχει αναπτυχθεί και έχουμε και την συμφωνία σύνδεσης ε, που θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, υλοποιηθεί και θα προκύψουν από εκεί θετικές εξελίξεις και ελπίζω μετά να οδηγηθούμε σε περαιτέρω μέτρα. κύριος Κριστέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε, Επίτροπε, έχουμε πολλές ελπίδες από τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και στη Ρουμανία που παρακολουθούν online αυτή την ακρόαση. Θα ήθελα απλώς να μου πείτε για την Δημοκρατία της Μολδαβίας και επειδή πλέον ε, ε κυβερνάται από δημοκρατική κυβέρνηση η οποία στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις που ε, οδεύουν προς την ε, ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ελπίζουν στη χώρα αυτή ότι κάποτε θα έχουν προοπτικές για προσχώρηση, για καθεστώς υποψήφιας χώρας. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο και ακόμη στρατηγική για την Μαύρη Θάλασσα, για τον Εύξενο Πόντο. Είναι κάτι που σας έχει απασχολήσει λόγω της, ε, των χωρών που βρέχονται από τη θάλασσα αυτή και του σφαιρικού της χαρακτήρα και για να προθεθούν όλα τα συμφέροντά μας σε αυτή την περιοχή. Ε, Τελευταίο που είπετε, ε, είπατε είναι ένα αναγκαίο συμπληρωματικό μέτρο και αυτή τη στιγμή το συζητούμε ε, με την είπατε εκπρόσωπο θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ασφαλώς και για τη Μολδαβία ισχύει το ίδιο όπως και για τις άλλες χώρες όπου ο πληθυσμός ε, ε, έκανε, δήλωσε ξεκάθαρα ότι θέλει να προσεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι θα πρέπει να το στηρίξουμε, να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Μολδαβία είναι η πρώτη χώρα με ένα καθεστώς απαλλαγμένο από την υποχρέωση θεώρησης ε, εισόδου. Ε, δεν, υπάρχει, δεν ισχύει η βίζα πλέον. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά είναι μέτρα στη κατεύθυνση. Και η Ρώμη δεν φτιάχτηκε σε μία μέρα και το ίδιο ισχύει για την προσέγγιση των διαφόρων χωρών προς την Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει το ένα βήμα να ακολουθεί το άλλο και θα πρέπει να επιδεικνύει κανείς την αναγκαία συνέπεια. Ε, θεωρώ ότι ε, οι εκλογές είναι ένα αναγκαίο βήμα και αν η έκβαση είναι θετική εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην υποστηρίξουμε περαιτέρω αυτή τη θετική εξέλιξη. Ω τελευταίο ομιλητή από τη δική μου πολιτική ομάδα, θα ήθελα να επιμείνω στα σημεία που δεν σα καταλάβαμε πολύ καλά. Πρώτον, τι σημαίνει reshaping, αναδιαμόρφωση της πολιτικής γειτονίας. Ε, ε, μετά από τρία χρόνια τι θα γίνει μετά από τρία χρόνια. Ε, παρουσιάσατε ότι είπατε ότι αυτό το οποίο εσείς δώσατε γραπτά και το... αυτό το οποίο δήλωσε ο κύριος Γιούνκερ ε, δεν, ε, δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί έτσι όπως ακούστηκε τελικά ότι θα υπάρξει μια συνέχιση διαπραγματεύσεων για παράδειγμα με χώρες όπως η Αλβανία, η οποία επιθυμεί την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων ή το Κόσοβο που δεν υπάρχει η ευκταία ρύθμιση για τη θεώρηση εισόδου. Τελευταία ερώτηση αφορά τη συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο. Θα ήθελα να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί θα θέλαμε να είστε ένας ισχυρός ε, επίτροπος και όχι απλώς παρατηρητής όταν το διακύβευμα είναι η Κύπρος η, η Μεσόγειος, επί παραδείγματι. Ε, απάντηση. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτά τα οποία έπρεξε μέχρι τώρα ο Στέφαν Φούλε ε, πραγματικά χρήσουν της δικής μας αναγνώρισης. Ε, δεν είναι εύκολο να σημειωθούν παραπέρα πρόοδοι. Ε, ε, και υπάρχει μια συνεργασία για θέματα, για περιπτώσεις όπως είναι η Αλβανία. Αλλά και ο κύριος ε, Φίλε ε, χρειάστηκε να περάσει μια περίοδο δοκιμής για να σκεφτεί πώς θα συνεχίσει. Εγώ είχα μέχρι στιγμής ε, μία εμπειρία στο επίπεδο των περιφερειακών ή ε, της διασυνοριακής ε, συνεργασίας και ο κύριος Γιούγκερ με παρακάλεσε τώρα στο νέο μου χαρτοφυλάκιο να συμπεριλάβω την πείρα αυτή που απέκτησα από την περιφερειακή πολιτική. Και Νομίζω ότι κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να δούμε την ε, λεγόμενη αναδιαμόρφωση πολιτικής γειτονίας, το reshaping. Και το ίδιο ισχύει και για την πολιτική της γειτονίας. Θεωρώ ότι πάρα πολλά μπορούν να επιτευχθούν με πολύ συγκεκριμένα προγράμματα, ειδικά όταν μιλάμε για τον Νότο, που θα πρέπει να ληφθούν πολλά ε, συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Και εδώ βλέπω ακριβώς το έβρος της συνεργασίας με την ε, κυρία Μοργκερίνη. Δηλαδή να, σε ε, η πολιτική μας με συγκεκριμένες ε, δράσεις. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις με την κυρία Μογκερίνη και νομίζω ότι το σκεπτικό μας είναι ότι θα πρέπει τα εργαλεία μας να εξυπηρετούν ε, τους στόχους της πολιτικής που έχουμε χαράξει. Γιατί ε, θα πρέπει και να μπορούμε να το στηρίξουμε ε, εμείς ήδη. Θα θυμάστε ότι ο κάθε επίτροπος έχει ένα δικαίωμα ψήφου στο σώμα των επιτρόπων και ε, όλοι θα συμμετάσχουν στην ε, διαμόρφωση της ε, περιφερειακής πολιτικής. Τώρα, όσον αφορά την Αλβανία, θα γίνει αυτή η έκθεση screening και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα ακολουθήσει τις δικές μας προτάσεις και θα πάρουν σχετικές αποφάσεις. Τώρα, για το Κόσοβο ε, ενημερώθηκα και μου είπαν ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν ακόμα κάποια τεχνικά ζητήματα και ελπίζω ότι μετά το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης θα βελτιωθεί η κατάσταση. Η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια έχει επιβάλει σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία και από την άλλη έχει κάνει επενδύσεις 120 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία αλλά και η Τουρκία κατάφορα παραβιάζει το διεθνή νόμο κατέχοντας στρατιωτικά εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει διαπράξει το έγκλημα της εθνοκάθαρσης σε βαθμό που στα κατεχόμενα εδάφη δεν υπάρχουν για γηγενείς ελληνικοί και χριστιανικοί πληθυσμοί, απειλεί συνεχώ την Κύπρο, δεν την αναγνωρίζει και την θεωρεί εγκλυπούσα σε επίσημα έγγραφα που καταθέτει στο Συμβούλιο. Πιστεύετε κύριε Επίτροπε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι συμβατή με συμπεριφορά κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείται σωστή την πολιτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών. Αυτή η πολιτική αυξάνει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς θα στηρίξετε έμπρακτα το πλέον αδύνατο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την επιθετικότητα ενός στρατηγικού εταίρου της Ένωσης. Σας ευχαριστώ oft diskutiert. Es ist auch wichtig, dass wir... Ναι. Κοιτάξτε, σημαντικό είναι εδώ πέρα να συνομιλούμε με όλους uh, τους ενδιαφερομένους. Εγώ γνωρίζω ήδη την κατάσταση στην Κύπρο αρκετά καλά. Είχα την ευχαρίστηση να συνομιλήσω και να συνεργαστώ με την Κυπριακή Προεδρία. Γνωρίζω, όπως είπα, την κατάσταση επιτόπου και Έχω ασχοληθεί και με έργα στην Τουρκία. Οπότε η τωρινή κατάσταση δεν είναι αποδεκτή και αυτό είναι ο λόγος ε, για τον οποίο δεν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Κρατών. Και οπωσδήποτε είναι θέμα το οποίο είναι συνεχώς πρώτο πρώτο στην ατζέντα το διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Κύριο Τζιπ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, είστε ένας από τους 7 επιτρόπους που ήσασταν και στην προηγούμενη επιτροπή και έχετε αρκετά μεγάλη εμπειρία από την περιφερειακή πολιτική. Θα ε, ήθελα να σα ρωτήσω ποιες από τι προηγούμενε εμπειρίες σας μπορείτε να μεταφέρετε στην πολιτική γειτονία. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών ή των οικονομικών επιχειρήσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τα ε, όργανα εξωτερικής χρηματοδότησης Ένωσης για αυτό τον σκοπό. Θα ήθελα να δω επίσης πώς σκοπεύετε να συμβιβάσετε τους πολιτικούς μας στόχους με τα μέσα, τα οικονομικά που έχετε στη διάθεσή σας. Κοιτάξτε, η εμπειρία μου ειδικά στον προγραμματισμό, την εφαρμογή, την εκτέλεση έργων μπορεί να φανεί χρήσιμη. Νομίζω πως ε, ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν ε, τον πρόεδρο Γιούνκερ να με προτείνει για αυτή τη θέση. Και στο πλαίσιο αυτό, αν μου δώσετε την εντολή, θα προσπαθήσω μέσω πολύ συγκεκριμένων ε, απτών ε, έργων να προωθήσουμε την ανάπτυξη αυτών των χωρών θα φροντίσω ιδιαίτερα ακριβώς να αυξηθεί το, η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις ε, υποψήφιες χώρες και στην γειτονιά μας. Γιατί με ενοχλούσε ως παρατηρητή το ότι δίνουμε τα περισσότερα λεφτά αλλά εμφανίζονται διάφοροι ε, οργανισμοί και οι άνθρωποι επιτόπου δεν ξέρουν τελικά πως ε, εκεί πέρα χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό ακριβώς ε, με ενδιαφέρει να φαίνεται δηλαδή ε, ότι τα λεφτά που πάνε κάπου είναι ευρωπαϊκά. Και νομίζω και αυτό συνεισφέρει στην επίτευξη των πολιτικών μας στόχων. Η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ανατέθηκε αυτό το χαρτοφυλάκιο, κύριε Χάν, και οι περισσότεροι στόχοι της εξωτερικής μας πολιτικής ακριβώς συμπίπτουν με το δικό σας πεδίο αρμοδιοτήτων. Εσείς μιλήσατε για τον διάδρομο Αδριατικής και Ιωνίου Πελάγος και τη διασύνδεση της δικής μας περιοχής με τους διαδρόμους TNT. Ε, είναι δύσκολο βεβαίως να προβλέψετε πόσο καιρό θα πάρει η οικοδόμηση του διαδρόμου Αδριατικής Ιωνίου Πελάγους, αλλά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και για τη Ποσνία Ερζεγοβίνη. Ε, ελπίζω αυτό που είπατε για την ποιότητα και την ταχύτητα να εφαρμοστεί και εδώ, όμως στη Βοσνία Ερζεγοβίνη τι και θα μπορούσαμε να δώσουμε στην προσχώρηση της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και μετά από μια πενταετία και μετά για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Χωρίς να αποθαρρύνουμε την Ουκρανία, πώς θα μπορούσαμε να τις, διαμορφώσουμε τις χώρες μας αυτές. Και στην Κροατία με τις χιλιάδες αγνοουμένους τι ε, μέλλον μπορούμε να δώσουμε και στα αιτήματα των ε, όσων αναζητούν τους ανθρώπους τους. Σουκά. Ε, δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα στα όσα είπατε στο τέλος, γιατί πραγματικά είναι δική μας υποχρέωση. Και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη ε, υπάρχει επιτέλους μια σωστή συγκοινωνιακή σύνδεση ε, που είναι μια ένδειξη ότι η Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι τμήμα επιτέλους της ε, Ευρώπης και βεβαίως ε, μελλοντικά μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Θα πρέπει να συνδέουμε τους ανθρώπους μεταξύ τους και ε, στη βάση αυτή θα μπορέσουμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα πράγματα. Ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό στα Δυτικά Βαλκάνια με συγκεκριμένες ε, δράσεις να μπορέσουμε να έχουμε μια συμβολή τους ώστε να αναπτυχθεί η περιοχή αυτή και να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν οι διάφορες χώρες εκεί ε, προς μια ε, προοπτική προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, κατά πρώτον συγχαρητήρια για την ε, ε, θητεία σας και σας εύχομαι κάθε καλή τύχη. Θε, έχω κατανοήσει τα επιχειρήματα και τα δικά σας και του Πρόεδρου Γιούνκερ και θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαδικασίες, ε, οι διαπραγματεύσεις μάλλον προσχώρησης, χωρίς προοπτική όμως να υπάρξει ένταξη πριν από μια πενταετία. Είναι μια σαφής απόφαση της ε, Επιτροπής Γιούνκερ αυτή. Τι θα γίνει όμως με τη δημοκρατία της Μολδαβίας εφόσον ε, επιτύχει τους στόχους της, αυτά τα κριτήρια που κλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρεί μέσα στο 2014. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δικής σας θητείας θα αναβαθμίσετε στις ε, διαπραγματεύσεις ένταξης την δημοκρατία της Μολδαβίας αν δείξει ότι είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Και ασχέτως με την ε, κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται η Ουκρανία και η Γεωργία γίνεται να αντιμετωπιστούν αυτές οι τρεις χώρες ανεξαρτήτως χωρίς να είναι ένα πακέτο. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές τις εξελίξεις. Οπωσδήποτε από την κυρία κάθε χώρα την αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά, την στηρίζουμε, αλλά να το ξαναπώ, πρώτα απ' όλα είναι κυρίαρχη απόφαση της κάθε χώρας και του λαού της. Και νομίζω πως ε, στην Μολδαβία τώρα στις εκλογές θα φανεί ποια πορεία θα ακολουθήσουν. Δεν είναι ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, και εγώ θέλουμε έχουμε κάποιον απότερο στόχο. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε μια κατάσταση στην οποία εάν έχουμε μια νέα χώρα μέλος θα είναι από την πρώτη μέρα σε θέση να λειτουργεί κανονικά εντός της Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε τις εμπειρίες της Ρουμανίας με τα προβλήματα απορρόφησης των διαρθρωτικών κονδυλίων κτλ. Καλό θα είναι να μην περάσουν τέτοια τα μελλοντικά κράτη-μέλη και να είναι σωστή η προετοιμασία για να έχουμε και επιτυχία. Κύριε Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε υποψήφια επίτροπε, γιατί ακόμα και αν μέσα στην ερχόμενη πενταετία δεν υπάρξει ένταξη κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ε, περί διεύρυνσης θα πώς θα δοθούν μάλλον κίνητρα στις υποψήφιες χώρες για να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις για να συνεχίσουν αμύωτες τις προσπάθειες να εκπληρώσουν τα κριτήρια για το κράτος το δημοκρατικό πολίτευμα, τον σεβασμό των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ουκρανία, η Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο είναι τρεις περιπτώσεις χωρών όπου τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι μεγάλης σημασίας. Υπάρχει ουγγρική μειονότητα, ρουμανική, σερβική, βλαχική που ζητούν ανεξαρτησία. Πρέπει λοιπόν να τους διασφαλίσουμε την σταθερότητα αλλά και την ένταξή τους σε μια ε, εύρυθμα λειτουργώσα κοινωνία των πολιτών. Αυτά είναι προαπαιτήσει και προποθέσει για την ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνετε εσεί για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των εθνικών, αθηνοτικών μειονοτήτων. Είναι κομμάτι των διαπραγματεύσεών μας με αυτές τις ε, χώρες και είναι νομίζω και στο άρθρο 2 της συνθήκης της Λισαβόνας. Προστασία των μειονοτήτων και πρέπει να το σεβόμαστε και η εμπειρία δείχνει πως ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών ε, συνεισφέρει στη λειτουργία μιας ε, κοινωνίας. Και έτσι εγώ προσωπικά λυπάμαι για να μην πω πονώ όταν ε, πρέπει να πιέσουμε για τέτοια πράγματα γιατί έπρεπε να είναι αυτονόητα. Γιατί όπως είπα δεν είναι μόνο κάτι το οποίο πρέπει να γίνει αλλά συνεισφέρει και στην ευημερία μιας κοινωνίας. Και οπωσδήποτε όπου δεν ε, γίνεται κάτι τέτοιο πρέπει να συνεισφέρουμε και εμείς και ξανά σας διαβεβαιώ, ειδικά όσον αφορά τις υποψήφιες χώρες, θα δούμε το θέμα αυτό με σοβαρότητα και με τον ξεκάθαρο στόχο να προετοιμαστούμε έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος από την πρώτη μέρα να είναι πλήρες μέλος και η εμπειρία δείχνει πως αυτό είναι και προς το συμφέρον αυτής της χώρας και των ανθρώπων της. Οπότε το αποφασιστικό είναι το, το αποτέλεσμα, όχι τα, τα πέντε χρόνια. Νομίζω πως τα πέντε χρόνια αυτά θα έχουμε καταφέρει ένα μεγάλο βήμα πρόοδου και ελπίζω όλοι μαζί να είμαστε τελικά ικανοποιημένοι και τελικά αυτός ο δακτύλιος της φωτιάς να έχει σπάσει σε αρκετά σημεία. Αυτός είναι ο προσωπικός μου στόχος. Σας ευχαριστώ.